η συνεδρίαση, η διάσκεψη των Προέδρων που σήμερα είναι ανοιχτή για όλα τα μέλη ξεκινάει τώρα και θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Τίμερμαν, τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το Κοινοβούλιο προετοιμάζει την ε, ψηφοφορία για την νέα Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 115 και το παράρτημα 16 του κανονισμού. Ε, προς αυτό έχουμε τα, τους προτινόμενους ε, υποψήφιους τους οποίους ε, εξετάσαμε σε σχέση με τις ικανότητές τους ε, και την ε, ανεξαρτησία της σκέψης τους. Επίσης, οι γνώσεις τους για τον χαρτοφυλάκιο τους και οι δυνατότητες επικοινωνίας και αυτές πρέπει να αξιολογηθούν. Και προς αυτό θα εξυπηρετήσει η σημερινή ακρόαση, η οποία είναι και η τελευταία πριν από την αξιολόγηση που θα λάβει χώρα από τους Προέδρους των Επιτροπών. Ο κύριος Τίμεμανς θα προβεί σε μια εισαγωγική δήλωση κατά το μέγιστο 15 λεπτών. Κατόπιν ε, θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις προς τον κύριο Τίμερμανς, συνολικά 45 ερωτήσεις που θα υποβάλλετε εσείς αγαπητοί συνάδελφοι. Και για κάθε ερώτηση προβλέπετε κατά το μέγιστο ένα λεπτό. Ο κύριος ε, Τίμερμανς ε, για να απαντήσει θα έχει δύο λεπτά για κάθε ερώτηση. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να τηρήσετε το χρονοδιάγραμμα και ως προς τις ερωτήσεις παρακαλώ να εστιάζεστε σε σημαντικά θέματα. Αυτή λοιπόν η ακρόση μεταδίδεται ζωντανά ε, στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και άλλη μια τεχνικής φύσεως παρατήρηση. Κυρίες και κύριοι, με γνωρίζετε, ξέρω ότι είμαι ένας πολύ φιλικός ε, και προσινής άνθρωπος, καλός άνθρωπος θα έλεγα, εκτός όταν πρόκειται για την υπέρβαση του χρόνου μιλίας. Και αυτό ως προς αυτό σήμερα θα είμαι ιδιαίτερα αυστηρός γιατί αλλιώς δεν θα μπορεί ο κύριος Τίμερσμαν να έχει χρόνο για να απαντήσει. Που σημαίνει ότι μετά από 15 δευτερόλεπτα θα αρχίσουν ε, να ανάβουν τα φωτάκια και μετά από 60 δευτερόλεπτα θα σας ε, παίρνω το λόγο. Λυπάμαι που ε, πρέπει να σας το πω ευθύς εξ αρχής αλλά πραγματικά το εννοώ. Κύριε Τίμερμαν, εσείς έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας για κάθε ερώτηση. Σας παρακαλώ λοιπόν, λοιπόν να τηρήσετε κι εσείς ε, το χρόνο. Δεν ξέρω, φαντάζομαι κι εσείς μπροστά σας ε, θα βλέπετε αυτά τα δύο κόκκινα στεράκια που τα αναποσβήνουν και θα δείχνουν ότι τελειώνει ο χρόνος σας. Ε, έχετε άλλες ερωτήσεις παρακαλώ, παρακαλώ επί της διαδικασίας. Όχι από ό,τι βλέπω. Κύριε Τίμερμανς, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, είναι μεγάλη τιμή και ευχαρίστηση για μένα που βρίσκομαι εδώ σήμερα μετά από δέκα έντονες μέρες όπου η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία απέδειξε την αριστεία της. Εφόσον επιβεβαιωθώ θα είναι η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία δημιουργήθηκε και γεννήθηκε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πνεύμα συνεργασίας και πολιτικού διαλόγου. Το 2014 είναι ένα ειδικό, ένας ειδικός χρόνος για την Ευρώπη. Εκατό χρόνια πριν είχαμε την αρχή δύο αυτοκτονικών πολέμων. 70 χρόνια πριν είχαμε την αρχή της απελευθέρωσης της Δυτικής Ευρώπης στα πλαίσια αυτού που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Οι ομάδες των κρατών δεν αναζητούσαν την ασφάλεια και την ευημερία με την δύναμη και την κυριαρχία αλλά με την ειρήνη και την ασφάλεια χρειάστηκαν να περάσουν αρκετά χρόνια και μόνο πριν 25 χρόνια η ιδέα αυτή έγινε ε, προσιτή για όλους τους Ευρωπαίους. Όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου ε, σταμάτησε και η βία και η κυριαρχία που ε, είχαν γίνει η μάστιγα της Ανατολικής Ευρώπης το Ανατολή και Δύση έγιναν όπως είχε πει ο Βάκλαβ Χάβελ αυστηρά γεωγραφικοί προσδιορισμοί και όχι πολιτικοί ή και ηθικοί δεοντολογικοί. Η μεγαλύτερη κόρη μου γεννήθηκε το 1986 όταν το τέλος της ε, ευρωπαϊκής διέρεσης ήταν κάτι που δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς. Ο μεγαλύτερος γιος μου το 89 όταν το, αυτό που δεν πίστευε κανείς έγινε πραγματικότητα και ο νεότερος το 4, το 2004 όταν πλέον οι νέες 10 χώρες είχαν ήδη ενταχθεί στην Ένωση. Έχει σημασία να δούμε πού βρισκόμασταν όταν βλέπουμε ποια είναι τα προβλήματα και μη με παρεξηγείτε τα προβλήματα είναι σοβαρά. Εάν επιβεβαιωθεί η Επιτροπή Γιούνκερ πρέπει να είναι σοβαρή στην αντιμετώπιση τους και αυτή. Δεν ξεκινάμε όμως τόσο άσχημα όσο λέγουν ορισμένοι αρκετά συχνά. Η Ευρώπη ήταν ικανή να αλλάξει τις κοινωνίες. Η Ευρώπη απέφυγε την πολυδιάσπαση και τους οικονομικούς και νομισματικούς πολέμους και αντιμετώπισε και ε, την καταστροφή την οποία πολλοί επέσιαν στα πλαίσια της χειρότερης κρίσης μετά το 1930. Ε, υπάρχουν προβλήματα βέβαια και τα μέτρα είναι οδυνηρά για πολλά εκατομμύρια Ευρωπαίων που δεν έχουν δουλειά και δεν έχουν πολλές ευκαιρίες. Οι προκλήσεις είναι τεράστιες, πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές. Θα πρέπει σαν πολιτικοί εμείς ε, να διαβεβαιώσουμε τους εκλογείς μας ότι αξίζουμε να μας εμπιστεύονται και θα μπορέσουμε να τους ικανοποιήσουμε. Εφόσον μας επιβεβαιώσετε θα χρησιμοποιήσω όλη μου την ενέργεια και την εμπειρία για να υποστηρίξω τον υποψήφιο πρόεδρο Γιούνκερ έτσι ώστε να πετύχει ε, το πρόγραμμά του για απασχόληση, ανάπτυξη και δημοκρατική αλλαγή. Θα πρέπει να δείξουμε με πρακτικό τρόπο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και τα ευρωπαϊκά όργανα δεν είναι αυτοσκοπή αλλά εξυπηρετούν τους πολίτες και τα κράτη-μέλη. Αυτά που πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα κάνει γιατί μόνο αυτή μπορεί να τα κάνει και τα υπόλοιπα θα τα κάνουν τα κράτη καλύτερα από αυτήν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα πρέπει να συγκεντρώσει την, επιτροπή, την ε, προσοχή της εκεί όπου μπορεί να βοηθήσει. Οι κατευθυντήριες πολιτικές γραμμές του κυρίου Γιούνκερ, του υποψηφίου Προέδρου της Επιτροπής, θα υποστηριχθούν από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως επίσης και από τις στρατηγικές προσανατολιστικές γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου καλύτερες νομοθετικές ρυθμίσεις, σωστότερες και ισχυρότερες διοργανικές σχέσεις, είναι σεβασμός επίσης του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πράγματα απαραίτητα για να αρχίσουν τα πράγματα να βελτιώνονται. Να δούμε ποιες είναι τώρα οι κοινέ πολιτικές μας προτεραιότητες. Εάν με επιβεβαιώσετε από τις αρχές του επομένου έτους θα προτείνω στο σύνολο των επιτρόπων κάποιες προτάσεις ε, οι οποίες είναι σε εκκρεμότητα και καιρό και θα πρέπει να αποσυρθούν αφού τις συζητήσουμε μαζί σας. Μέσα σε ένα χρόνο θα παρουσιάσω μια ε, ε, μια επισκόπηση θα έλεγα των ε, βελτιώσεων στον τομέα της νομοθεσίας για να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τα συμφέροντα της Ευρώπης. Αν το πετύχουμε αυτό είμαι βέβαιος ότι θα γίνει μια σωστή πολιτική συζήτηση για τον πολιετή προγραμματισμό σύμφωνα με το άρθρο 17 της συνθήκης εφόσον μας επιβεβαιώσετε στη θέση αυτή. Θα βελτιώσουμε επίσης και το σύστημα αξιολόγησης των επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ενθαρρύνουμε το Συμβούλιο να ακολουθήσει την ηγετική θέση, την πρωτοπορία την οποία έχει επιδείξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι σαφές ότι οι αλλαγές που έχουν γίνει θα πρέπει να ληφθούν υπόψη βέβαια. Έχει μεγάλη σημασία και η Επιτροπή, ε, το Συμβούλιο μάλλον αξιολόγησης επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να δράσουν και να κρίνουν ανεξάρτητα. Εγώ θα εκφράζω την άποψή μου για τις εκθέσεις αυτές όταν παρουσιάζονται στην Επιτροπή και όταν χρησιμοποιείται μια κίτρινη ή πορτοκαλί κάρτα τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να το αντιμετωπίζει πολύ προσεκτικά, θα πρέπει η Επίτροπη να είναι σε στενότερο διάλογο με τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Εφόσον με εγκρίνεται, ρόλος μου θα είναι να ενθαρρύνω τους συναδέλφους μου να συζητούν άμεσα με τα κοινοβούλια των κρατών μελών και να ακούν τις απαντήσεις και τις ερωτήσεις και να δίδουν και απαντήσεις. Τα αποτελέσματα αυτών των συζητήσεων θα πρέπει να τα μοιραζόμαστε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να καταλάβουμε όλοι πραγματικά τι σημαίνει επικουρικότητα, κάτι που θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφύγει τις μη απαραίτητε προτάσεις, έτσι ώστε να υπάρχει βέλτιστη δυνατή παρέμβαση όπου αυτό είναι απαραίτητο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινότητα εθνών και πολιτών οποίοι τις τελευταίες δεκαετίες ήρθαν κοντά ο ένας τον άλλο χωρίς να αμφισβητήσουν ποτέ την εθνική τους ταυτότητα ή τη σημασία των κρατών εθνών. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι ισχυρή μόνο αν τα κράτη-μέλη είναι ισχυρά και η ισχύ ε, ε, των κρατών μελών εξαρτάται και από την ισχύ της Ένωσης. Η προσωπική μου εμπειρία μου λέγει ότι μόνο από κοινού θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε θέματα σφαιρικά όπως οι κλιματολογικές αλλαγές, η τρομοκρατία και να αντιμετωπίσουμε ε, με θετικό τρόπο τις επιλογές κυριαρχίας και ανεξαρτησίας χωρών όπως η Ουκρανία. Κράτη λοιπόν και πολίτες είναι τα βασικά συστατικά της Ένωσης. Θα αποτύχουμε αν δεν λάβουμε υπόψη μας και τα δύο αυτά στοιχεία. Είναι στη φύση των πολιτικών σωμάτων να δώσουν περισσότερη προσοχή σε νέες πρωτοβουλίες και στην αξιολόγηση της υπάρχουσας νομοθεσίας. Θα πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Απαιτείται να γίνουμε καλύτεροι ακούγοντας τους πολίτες μας και τις επιχειρήσεις οι οποίοι είναι αυτοί που εφαρμόζουν την νομοθεσία και θα πρέπει να είμαστε απολύτως βία ειλικρινείς θα έλεγα όταν περιγράφουμε το τι δεν πάει καλά και πρέπει να αλλάξει ή όπου έπου έχουμε αποτύχει. Θα πρέπει λοιπόν οι εμπλεκόμενοι όχι απλά να τους συμβουλευόμεθα εδώ στις Βρυξέλλες αλλά να εκπροσωπούνται σωστά εδώ στις Βρυξέλλες. Απαιτείται μεγαλύτερη επίσης διαφάνεια. Γι' αυτό θα προωθήσω και μια διοργανική συμφωνία για ένα υποχρεωτικό κατάλογο των καταγεγραμμένων λόμπις. Ε, δεν μιλάμε για έλλειψη νομοθεσίας, ε, για απελευθέρωση στον τομέα το διακανονιστικό, όχι, μιλάμε για μείωση της γραφειοκρατίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να δημιουργούνται νέες επιχειρήσεις, να δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης ε, και να αποφεύγονται απαράδεκτες και μη χρήσιμες νομοθετικές ρυθμίσεις. Θα αποτύχει η προσπάθειά μας αν επιτίθεται στα κοινωνικά δικαιώματα και την περιβαλλοντική προστασία. Εάν πράγματι θέλουμε εμείς να γίνουμε καλύτεροι νομοθετικά τότε θα έρθουμε σε στενότερη επαφή με τους εμπλεκόμενους οι οποίοι απογοητεύονται γιατί πιστεύουν ότι η Ευρώπη είναι η πηγή της γραφειοκρατίας. Εγώ δεν είδε ολυπτό σε σχέση με αυτό. Προσπαθώ να σκεφτώ πρακτικά και προσπαθώ να είμαι και επιλεκτικός εκεί που χρειάζεται. Εφόσον με επιβεβαιώσετε στη θέση μου θα στηρίξω τους συναδέλφους μου ε, στις σωστές τους επιλογές και θα σημειώσω τη διαφωνία μου με τις μη σωστές επιλογές. Γιατί ο κόσμος μας βλέπει όλους σαν ένα πράγμα. Λένε ποιοι, α οι Βρυξέλλες, πηγή απογοήτευσης ανεξάρτητα από τις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε. Κατηγορώντας τα άλλα κοινοτικά όργανα δεν είναι κάτι που βοηθάει. Εμείς θα πετύχουμε μόνο αν από κοινού πολεμήσουμε και για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να αλλάξουμε γιατί αλλιώς ε, δεν ε, θα δείξουμε ότι καταλαβαίνουμε το πόσο κατεπίοντα είναι τα προβλήματα. Θα σεβαστούμε βέβαια τις ευρωπαϊκές αξίες και τις αρχές μας, αυτά που μας ενώνουν μέσα στη διαφορετικότητά μας θα είμαστε επίμονοι στην εφαρμογή του νόμου από τα ευρωπαϊκά όργανα και από όλα τα κράτη-μέλη. Αν αποτύχει ένας από εμά επηρεάζεται και θίγεται η αξιοπιστία όλων μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεματοφύλακας της συνθήκης και της Χάρτας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι υπεύθυνη για την σωστή εφαρμογή τους. Θα είναι προσωπική μου ευθύνη ε, το να δώσω ε, επίσης προτεραιότητα σε αυτήν την συγκεκριμένη αρμοδιότητα την τόσο σημαντική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διαβεβαίωση λοιπόν του σεβασμού και της εφαρμογής του κράτους δικαίου και του νόμου μαζί με τους συναδέλφους στο σύνολό τους. Και όταν πάρουμε την γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα πάρουμε τα απαιτούμενα βήματα έτσι ώστε να δούμε τι θα γίνει και σε σχέση με τη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, θα συνεργαστώ με όλες τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις που έχουν σαν στόχο την προώθηση και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η επιτυχία του ενός είναι επιτυχία όλων, γιατί όλοι συμμεριζόμεστα Όλοι συμμεριζόμαστε έλεγα τα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδη δικαιώματα. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για μεγαλύτερη πολιτική εμπλοκή στον τομέα αυτό όπως έχετε και εσείς υπογραμμίσει. Θα οργανώσω ένα ετήσιο συνέδριο για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη με την πλήρη συμμετοχή όλων των θεσμικών οργάνων, των σχετικών όπως και του Κοινοβουλίου προφανώς. Αγαπητά μέλη, κυρίες και κύριοι. Εισαγωγικά σας μετέφερα κάποιες σκέψεις γιατί τα θέματα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά εφόσον με επιβεβαιώσετε στη θέση αυτή. Θεμελιώδη δικαιώματα, καλύτερη νομοθετική ρύθμιση και μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υπηρετεί τους Ευρωπαίους. Φυσικά ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός. Είμαι στη διάθεσή σας για να σας ακούσω, να δεχθώ τις ερωτήσεις σας και να ξεκινήσει ένας πραγματικός πολιτικός διάλογος. Αυτά που προτείνουμε δεν είναι εύκολα και δεν είναι κάτι το δεδομένο. Οι αλλαγές είναι δύσκολες. Ο τρόπος με τον οποίο έχουμε οργανωθεί. Η μία αλλαγή όμως ε, θα είναι κάτι το πάρα πολύ πιο οδυνηρό. Η αλλαγή την οποία προτείνει η Επιτροπή Γιούνκερ είναι θεμελιώδης αν θέλουμε πράγματι να αναπτυχθεί και να ξανάρθει η ελπίδα στην Ευρώπη. Αν θέλουμε να πετύχουμε δεν θέλουμε μόνο την στήριξή σας αλλά την πλήρη εμπλοκή σας. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και μερικές φορές μπορεί να απογοητευτούμε. Αλλά όμως μία από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι παππούδες μας και οι γονείς μας <clears throat> είναι ότι τα κατάφεραν και φυσικά η Ευρώπη έχει περάσει από πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις και κατάφερε και συνήλθε. Πρέπει λοιπόν να εξυγχρονίσουμε ε, και να βελτιώσουμε την Ευρώπη σήμερα. Έτσι ώστε η κληρονομιά των πατέρων της Ευρώπης να μην χαθεί στα βιβλία της ιστορίας. Αυτή είναι η Ευρώπη την οποία θέλουμε και είμαστε συλλογικά υπεύθυνοι για αυτήν. Είναι δύσκολη αυτή η προσπάθεια, αλλά ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα αποδείξουμε ότι είμαστε ικανοί. Ας καταστήσουμε τους πατέρες μας περήφανος, ας καταστήσουμε τα παιδιά μας περήφανα και ας επιτρέψουμε στην Ευρώπη να στοχεύσει και να επιστρέψει σε ένα λαμπρότερο μέλλον. Das Wort hat Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τιμερμάν. Στο λόγο έχει ο κύριος Γκοντσάλης Πόντς. Παρακαλώ. Να σας καλωσορίσω εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κύριε Τίμερμαν. Θα ήθελα καταρχάς να σας πω ότι συμμεριζόμεθα τις αξίες τις οποίες αναφέρατε στην προηγούμενη παρουσία σας. Εμείς πράγματι θέλουμε να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες, την, αξιο, την αξιοπρέπεια, την προσωπική, την αλληλεγγύη. Είναι θα έλεγα κομβική τομή της προσπάθειας την οποία θα πρέπει να κάνουμε. Η προστασία αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, θα μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε και την τρομοκρατία και το, το οργανωμένο έγκλημα στα πλαίσια πάντα των νόμων του κράτους δικαίου. Έτσι θα υπερασπιστούμε τον χώρο της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, το οποίο θέλουμε να είναι και να συνεχίσει να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην παρούσα φάση και στο Ιράκ και στη Συρία υπάρχουν ε, εκατοντάδες Ευρωπαίοι δυστυχώς οι οποίοι ασκούν τρομοκρατικές δραστηριότητες και είναι έτοιμοι να σκοτώσουν. Λοιπόν η πρώτη μου ερώτηση είναι εξής. <clears throat> Τι συγκεκριμένα μέτρα θα πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προστατεύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους Ευρωπαίους πολίτες από την τρομοκρατία. Thank um, Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Πρόκειται για ένα από τα πιο ακαθόδη θέματα. Τα έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό σήμερα. Και προκαλεί έκπληξη ότι κάποιοι από τους πλέον ευφυείς ε, νέους ανθρώπους στις χώρες μας μπαίνουν στον πειρασμό να πάνε σε άλλες χώρες και να πολεμήσουν και να καταπολεμήσουν μάλιστα τις πιο θεμελιώδεις αξίες τις οποίες έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά να επανέλθουν για να απειλήσουν άμεσα την κοινωνία μας. Είναι αυτονόητο ότι οι κοινωνίε έχουν το δικαίωμα να προστατευτούν, να αυτοπροστατευτούν κατά της τρομοκρατία αυτής και θα πρέπει να συνεργαστούμε ω έθνη πιο στενά για να εξασφαλίσουμε ότι θα δώσουμε απάντηση σε αυτή την άμεση απειλή για την ασφάλειά μας. Πρόκειται για ένα, σαφ... για σαφή κίνδυνο για την ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων. Πρόκειται για μια ευθύνη πρωτευόντως των κρατών μελών, προφανώς αλλά σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν μπορεί να μας επιτρέψει να αμελήσουμε τα ίδια τα θεμελιώδη δικαιώματα που θέλουμε να προασπίσουμε. Στην καταπολέμηση λοιπόν της τρομοκρατίας θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν περιορίζουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των πολιτών μας. Γιατί αν το κάνουμε αυτό, αν κάνουμε τέτοιο συμβιβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα, θα βλάπταμε ουσιαστικά τις ίδιες αξίες που καταπολεμούν αυτοί οι τρομοκράτες. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι κάθε ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο και κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τηρεί τις αρχές που κατοχυρώνονται στον χάρτη και στην συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα εξ ονόματος ε, της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του οποίου με θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω για την πάρα πολύ καλή εισαγωγή που κάνατε κύριε Αντιπρόεδρε. Κατά τις τελευταίες εκλογές ε, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα στους πολίτες και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Υπάρχει το ευρωπαϊκό εγχείρημα το οποίο δυστυχώς απειλείται και το αντίδοτο σε αυτή την κατάσταση θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών πολιτών. Η Κομισιόν θα πρέπει λοιπόν να αντιστρέψει την πυραμίδα, οι αποφάσεις να μην είναι απαραίτητα από πάνω προς τα κάτω, αλλά να υπάρχει συμμετοχή. Και στο, στη συνθήκη της Λιβόνας υπάρχει ένα εργαλείο. Είναι το δικαίωμα των πολιτών να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για πάρα πολλά θέματα. Για το περιβάλλον, για την εργασία, για τον υδροφόρο ορίζοντα. Αυτό λοιπόν είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο το οποίο έχουμε στα χέρια μας. Εσείς λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω πώς ακριβώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε αυτή την απειλή η νέα επιτροπή. Πώς θα συμβάλλει έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί το δημοκρατικό οικοδόμημα. Κοιτάξτε, εγώ ίδιος ανέλαβα την πρωτοβουλία κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Υπάρχει αυτό αυτή πρωτοβουλία, το δικαίωμα αυτό των πολιτών και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το οποίο βιώσαμε τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή δηλαδή αντιδρούσε με έναν τρόπο που τον κατανοώ πάρα πολύ καλά, όμως μερικές φορές αυτός ο τρόπος ήταν πάρα πολύ νομικίστικος, στεγνός και η ε, αντίδραση των πολιτών ε, δεν είναι σε σχέση με αυτή τη στική στάση, αλλά την πραγματικότητα. Δηλαδή να υπάρχει μια περισσότερο πολιτική στάση της Επιτροπής οποτεδήποτε λαμβάνονται πρωτοβουλίες εκ μέρους των πολιτών. Είναι απαραίτητο η Επιτροπή να θεωρεί ότι αυτές οι πρωτοβουλίες είναι πολιτικής φύσεως. Βεβαίως καταλαβαίνω αυτά που αναφέρει η συνθήκη και προφανώς οφείλουμε να σεβόμαστε τη συνθήκη γιατί η συνθήκη μας κατευθύνει. Αυτό όμως όμως μας προσφέρει και τη δυνατότητα να έχουμε και πολιτική συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα. Όταν οι πολίτες αισθάνονται ανασφάλεια για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Κομισιόν ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι πολίτες επιθυμούν πολιτική συζήτηση, ε, τότε ας επιτύχουμε μια συμφωνία ανάμεσα σε Κοινοβούλιο και Κομισιόν να αναζητήσουμε τη συζήτηση με τους πολίτες και όχι μόνο με αυτούς που εκπροσωπούνται εδώ στις Βρυξέλλες, αλλά με εκείνους τους πολίτες που βρίσκονται στα κράτη-μέλη επιτόπου που θέλουν να βλέπουν κοντά τους επιτρόπους και κοντά τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βαντάλεν παρακαλώ. πολύ πολίτες είναι επικριτική κατά της Ευρώπης και αυτό το βλέπουμε στις προσέλευσεις στις ευρωπαϊκές εκλογές και στην χαμηλή, στα χαμηλότερα ποσοστά και στις επιχειρήσεις δεν είναι τόσο αγαπητή η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός και αν πρόκειται για επιδοτήσεις, γιατί συχνά μας λένε ότι μας επιβάλλει πάρα πολλούς κανόνες η Ευρώπη. Πώς μπορεί λοιπόν να περάσει ο Επίτροπος για την καλύτερη νομοθεσία ε, την Ευρώπη από τον εκνευρισμό στην ικανοποίηση. Είπατε ότι θέλετε να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά η Ευρώπη, πιο αποδοτικά. σε ό,τι αφορά τα όρια των 34.000 ευρώ για τα ενίκη, για παράδειγμα, και άλλα ενοχλητικά μέτρα. Λοιπόν, πείτε μου συγκεκριμένα ποια μέτρα θα λάβετε για να περάσει λοιπόν η Ευρώπη από τον εκνευρισμό σε, και να καταστεί σημείο φιλοδοξία πραγματικά και έμπνευση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σα, ο κύριο Τίμερμαν. Αν ήσασταν ε, πέρσι μαζί μου στο Κίεβο την ίδια εποχή, θα Βλέπατε πώς εμπνέει η Ευρώπη ακόμα. Η Ευρώπη για πολλά εκατομμύρια Ευρωπαίους αποτελεί πηγή έμπνευση και ένα φράγμα, αν θέλετε, σε έναν κόσμο με πολλές ανασφάλειες. Δεν υπάρχει λοιπόν έλλειψη για... σε ό,τι αφορά την έμπνευση. Αλλά έχετε δίκιο. Ενοχλεί και η Ευρώπη και έχει σημαντικά ελαττώματα, ελλείμματα σε ό,τι αφορά την νομοθεσία, την εφαρμογή της νομοθεσίας και όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα χτενίσουμε. Χρειάζομαι το κοινοβούλιο σας γι' αυτό. Θα το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχω προεξαγγείλει κάποια μέτρα, αλλά χρειάζομαι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω και το Κοινοβούλιο να πάρει πολύ στα σοβαρά τη μελέτη αντικτύπου που έχει ε, εξαγγείλει και θέλω μαζί να πείσουμε το Συμβούλιο και αυτό να κάνει η μελέτη αντικτύπου για το τι θα πρέπει να αλλάξει. Και θα ήθελα αυτά να γίνουν βράχοι πρόθεσμα. Όλοι οι μικρομεσαίοι, όλοι οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι που τώρα, αν τους ρωτούσαμε τι θεωρείς για την Ευρώπη και μας θα λέγανε «Α, με ενοχλεί». Σύντομα λοιπόν να λάβουν ένα περιθώριο προκειμένου να μπορέσουν να προσλάβουν καινούργια άτομα, να έχουν πιο πολλή επιχειρηματικότητα. Για παράδειγμα, στους φούρνους, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Γιατί η χώρα που γνωρίζω πιο καλά από όλες, έκανε μια σχετική οικονομική ανάλυση. Βλέπουμε λοιπόν ότι για τις μικρές επιχειρήσεις, ακόμα και μια μικρή μείωση της γραφειοκρατίας θα σήμαινε δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον ατόμων. Τι χρειάζεται λοιπόν η Ευρώπη στα μικρομεσαίο επίπεδο, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πιο πολλέ θέσει απασχόληση. Για το 85% των εργαζομένων απασχολείται σε αυτό το κλάδο. Αυτό λοιπόν πιστεύω θα επιφέρει αποτελέσματα. Η κυρία Ιντφέλντ, ευχαριστώ. Κύριε Τίμερμαντ. Η ομάδα του Άλντε καλωσορίζει τη νέα καινοτομική Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τους αντιπροέδρους της. Ωστόσο, κάποιοι υποψήφοι δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν το νεοδητό σύστημα. Τι μέσα λοιπόν έχετε, τι δυνατότητες και εξουσίες έχετε ως πρώτος αντιπρόεδρος για να πειθαρχήσετε τους άλλους ε, επιτρόπους και αν δεν υπάρχουν πραγματικά τέτοιες αρμοδιότητες, μήπως είναι εκ των προτεραιών νεκρό αυτό το σύστημα. Κατά δεύτερον, για την ΑΛΔΕ, οι ευρωπαϊκές αξίες είναι τη σημασία, όπως και για εσάς φαντάζομαι. Και θα πρέπει λοιπόν εν ώψη των φανατικών στην Ευρώπη να αντιδράσουμε προκειμένου να καταστήσουμε τη δημοκρατία μας πιο στεναρή. Είπατε ότι θα ε, ενισχύσετε τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά προσθέτετε και μία δήλωση ότι θα λαμβάνονται υπόψη αυτή η θεσμική και πολιτισμική ε, ποικιλομορφία της Ευρώπης. Τι σημαίνει αυτό ότι θα εθροτυφλήσετε, ότι θα γυρίσετε την πλάτη σε περίπτωση που καταπατώνται διάφορα θεμελιώδη δικαιώματα στα, στο όνομα της ε, εθνικής πολυμορφίας. Θα είσαστε λοιπόν πρωταθλητής των δικαιωμάτων τι θα είσαστε ακριβώς, ο κύριος Τίμερμανς ε, απάντηση. Πολύ καλή ερώτησή σας, κυρία Εντφέλτ. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τη δεύτερη ερώτηση, γιατί θεωρώ ότι είναι ουσιώδες το θέμα. Νομίζω ότι θα προσπαθήσω να συνεργαστώ με όλους στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την πρόθεση των θεμελιδών δικαιωμάτων. Θέλω να δημιουργήσω ένα δίκτυο θεσμικών οργάνων που θα ενισχύουν το ένα το άλλο και να συνεργαστώ στενά με το Συμβούλιο τη Ευρώπη με το, την οργάνωση των θεμελιωδών δικαιώματα, με την Επιτροπή της Βενετίας και με τους ακτιβιστές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πλαίσια ΜΚΟ. Και σίγουρα δεν πρόκειται να κάνω εκπτώσεις σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δεν υπάρχει καμία πολιτισμική δικαιολογία, κανένα πολιτισμικό πλαίσιο που θα δικαιολογούσε κατά καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προσυπογράψει τη χάρτα που έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από όλα τα κράτη-μέλη. Το μόνο που μπορώ να κάνω λοιπόν είναι να καλά τα κράτη-μέλη να τηρούν και να εκπληρούν τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει και θα χρησιμοποιήσω οποιοδήποτε μέσο έχει στη διάθεση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εφαρμόσω τις ιδέες αυτές, αυτούς τους κανόνες τους οποίους τα κράτη-μέλη έχουν προσυπογράψει σε ό,τι αφορά την σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επικεντρωθεί στις προτεραιότητες που όρισε ο υποψήφιος πρόεδρος Γιούγκερ και που ο πρόεδρος Γιούγκερ και που αποφάσισε το Κοινοβούλιο. Θα διασφαλίσουμε ότι η σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μας επιτρέψει να επικεντρωθούμε στα πρωτεύοντα ζητήματα και προφανώς η συνθήκη αποτελεί τη βάση, η συνθήκη αποτελεί τη βάση της εντολής του κάθε επιτρόπου και επίσης δίνει το δικαίωμα στον πρόεδρο να οργανώσει την επιτροπή του και ο πρόεδρος Γιούγκερ το έπραξε αυτό με τρόπο που θα μας επιτρέψει να επικεντρωθούμε στις προτεραιότητες μας και θα αποδείξουμε ότι μπορούμε λοιπόν να το πετύχουμε. Η κυρία Τσίμε, Κύριε Τίμεμανς, ε, από ό,τι κατάλαβα ε, δεν θέλετε να είσαστε ουραγός και ίσως ε, θα ήταν καλύτερα αντί για δεξί χέρι να γίνετε το αριστερό χέρι του κυρίου Γιούγκερ. Γιατί στην περίπτωση αυτή τότε θα μπορέσετε να υπερασπιστείτε τα δικαιώματα των πολιτών ε, και κυρίως και θέματα πολιτισμού. Αυτά να τα μεταφέρετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Τρόικα, οι πολιτικοί λιτότητα οδήγησαν σε παραβίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω πώς θα μπορέσετε να εμποδίσετε στο πλαίσιο της αξιολόγησης νομοθετικών πράξεων και πολιτικών να μην προκύπτουν παραβιάσεις θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι όσον αφορά το διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πώς θα μπορέσετε να βελτιώσετε τη συμμετοχή των κρατών μελών για τα μεγαλεπίβολα προγράμματα επενδύσεων, έτσι ώστε δηλαδή και τα κράτη-μέλη να διαθέτουν τα κονδύλια που τους αναλογούν. Όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, προφανώς και θα τα υπερασπιστούμε τόσο στα κράτη-μέλη όσο και στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φαντάζομαι, θα έχετε ακούσει, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Γιούγκερ, στην παρουσίασή του ανέφερε ότι θα μεριμνήσει έτσι ώστε στα μέτρα που θα ληφθούν να συμπεριλαμβάνεται και η κοινωνική διάσταση. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμπεριλαμβάνονται στον προγραμματισμό μας και οι συνέπειες, οι αξιολόγηση των συνεπειών μέτρων. Αυτό το έχει υποσχεθεί ο κύριος Γιούγκερ και νομίζω ότι θα το πράξει. Τώρα, όσον αφορά το διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια, νομίζω πρέπει να μεριμνήσουμε ε, για να κινητοποιηθούν κονδύλια, οπουδήποτε υπάρχουν αυτά, έτσι ώστε τα κονδύλια να μπορούν να επενδυθούν στην ευρωπαϊκή οικονομία, να υπάρξουν περισσότερες θέσεις απασχόλησης και να υπάρξει και πάλι μεγαλύτερη ελπίδα για τους Ευρωπαίους πολίτες που πραγματικά υπέφεραν πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της κρίσης. Και όπως υπενήχθηκε και ο κύριος Γιούγκερ, όλα αυτά σχετίζονται με το δικό μας τον προϋπολογισμό, με τους εθνικούς προϋπολογισμούς, με επενδύσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Αυτά έχουμε κατά νου και θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Γιατί, όπως είπε χθε και ο συνάδελφος Ντομπρόφσκι, Τώρα πλέον έχει φτάσει η στιγμή να γίνουν οι επενδύσεις στην Ευρώπη και είμαι πεπισμένος ότι εκεί θα τα καταφέρουμε. Ο κύριος Λαμπέρ αν μπορέσω να σας δώσω την ευκαιρία να μιλήσετε και γαλλικά κύριε Τίμερμανς. Εντάξει, ίσως ελεύθερα κάνω την εξής ερμηνεία ότι σε έναν κόσμο ο οποίος ε, ε, κυριαρχείται από την ανισότητα, ο νόμος είναι αυτός που μπορεί να μας επαναφέρει στην τάξη. Και γι' αυτό θέλω να μου δώσετε λεπτομέρειες για το better regulation, λέει στα αγγλικά ο κ. Λάμπερτς, ε, σε δύο σημεία μιλήσατε ότι δεν πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση της φορολογίας των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Βλέπετε όμως ότι ακριβώς επειδή έχουμε 26 διαφορετικά καθεστώτα, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις ελέγχουν ουσιαστικά την ζωή μας και όχι η ίδια η δημοκρατία. Ο μηχανισμός ISDS που θέλουμε να εντάξουμε στις εμπορικές συμφωνίες τώρα. Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο ε, δίνει κίνητρα στα κράτη ουσιαστικά για να μην νομοθετούν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αν θέλετε ο Πρόεδρος και εγώ μπορεί να μιλάμε και την τοπική μας διάλεκτο αλλά για την ε, εναρμόνιση τη φορολογική, το αίτημα. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν περιορισμοί στη συνθήκη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κάνει προτάσεις, αλλά οι προτάσεις αυτές βασίζονται στη συνθήκη, δεν μπορούν να βήγουν από τη συνθήκη. Εάν προτείνεται αλλαγές στο εσωτερικό της συνθήκης, αυτό θα το δούμε σε κάποια φάση. Οι προτάσεις μας θα ε, βασίζονται πάντα στη συνθήκη όσο έχει τουλάχιστον σήμερα και γι' αυτό ακριβώς δεν βλέπω να υπάρχει συγκεκριμένη αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα που αναφέρατε, της εναρμόνισης της φορολογίας. Τώρα για την πρόσβαση στα δικαστήρια, η συνάδελφος Γιώργοβα ήταν ξεκάθαρη σε σχέση με αυτό. Και νομίζω επίσης και άλλοι επίτροποι στους οποίους θέσατε τις ερωτήσεις αντίστοιχα. δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να περιοριστούν τα δικαιώματα ε, των Ευρωπαίων πολιτών για την προσφυγή τους στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Στην περίπτωση που υπάρχουν συγκρούσεις δικαιοδησιών κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι στα πλαίσια της συνθήκης που θα διαπραγματευτούμε δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να περιοριστεί η δυνατότητα πρόσβασης όσο έχει τουλάχιστον σήμερα. Στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν με διάφορες χώρες λοιπόν και με τις Ηνωμένε Πολιτείε είναι μια συγκεκριμένη δέσμευση αν θέλετε από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Μπορέλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εσείς είσαστε ε, υπεύθυνο για το Better Regulation και για τον συντονισμό των χαρτοφυλακίων της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Γνωρίζουμε και μας ανησυχεί άλλωστε αυτό ότι ένα σημαντικό τμήμα των κοινοτικών πιστώσεων καταλήγουν στα ταμεία του οργανωμένου εγκλήματος. Πώς σκοπεύετε εσείς να εργαστείτε και τι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σκοπεύετε να αναλάβετε στους τομείς αυτούς έτσι ώστε να σταματήσει πλέον η ροή κοινοτικών χρηματοδοτήσεων προς επιχειρήσεις και τοπικές αρχές οι οποίες καλύπτουν ε, και αρχές μάλλον που καλύπτουν ουσιαστικά τη δραστηριότητα του οργανωμένου εγκλήματος. Συνεχίζει ο κύριος Τίμερμαν Ιταλικά. Εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη ευθύνη από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παίρνουμε αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που επηρεάζουν άμεσα τα κράτη-μέλη. Ταυτόχρονα όμως και για τις πιστώσεις στις οποίες αναφερθήκατε κύριε Μπορέλη. Υπάρχει μια μεγάλη ευθύνη από πλευράς των κρατών μελών και πολύ συχνά υπάρχει και μια μεγάλη ευθύνη ε, υπηρεσιών αν θέλετε, οντοτήτων που δεν ανήκουν στην κεντρική κυβέρνηση αλλά στην περιφέρεια και σε άλλες μορφές οργάνωσης. Πρέπει λοιπόν εδώ να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμεθα με τα κράτη-μέλη, για να είμαστε βέβαιοι ότι οι πιστώσεις αυτές τίθενται στην διάθεση αυτών που τα, χρειάζονται, που τις χρειάζονται τις πιστώσεις αυτές. Αυτό ίσως το αφήνουμε πάρα πολλές φορές σαν ευθύνη στα κράτη-μέλη αποκλειστικά. Ενώ εδώ υπάρχει μια ευθύνη μεν των κρατών μελών αλλά και των ευρωπαϊκών οργάνων είναι υποχρέωσή μας προς τους Ευρωπαίους πολίτες που πληρώνουν τους φόρους αυτούς έτσι ώστε να δίνουμε εμείς τις ενισχύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους και σε συνεργασία με το ελεγκτικό συνέδριο για να είμαστε βέβαιοι ότι στο μέλλον να γνωρίζουμε καλύτερα το πού πηγαίνουν οι πιστώσεις αυτές ε, όταν διοχετεύονται στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφια Επιτροπέ, είπατε ότι την επόμενη χρονιά θα παρουσιάσετε τη θεσμική ε, συμφωνία για την καλύτερη νομοθεσία. Θα θυμάστε ίσως ότι το 2003 το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο αποφάσισαν να βελτιώσουν το συντονισμό ε, σε ό,τι αφορά την καλύτερη νομοθεσία και σε ό,τι αφορά τη συνθήκη στο άρθρο 17 για την ε, διάταξη για τον προγραμματισμό σε ό,τι αφορά την νομοθεσία. Δυστυχώς δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φαντάζομαι ότι οι πολίτες από εμά περιμένουν πιο αποτελεσματικό τρόπο δράσης. Και αν υπάρχει αυτή η νομοθετική, ο νομοθετικός προ, προγραμματισμός σε αυτό, το, σε αυτό το συντονισμό, θα α, τσακωνόμαστε λίγο λιγότερο και θα επικεντρωθούμε σε θέματα ουσίας. Ρωτώ λοιπόν, προγραμματίζεται μια εντελώς καινούργια τη θεσμική συμφωνία σε ό,τι αφορά το, τη συμπερίληψη του νομοθετικού προγραμματισμού. Θα βασιστείτε σε αυτή τη 2003, προσθέτοντα την διάσταση του νομοθετικού προγραμματισμού ή έχετε υπόψη κάτι εντελώς διαφορετικό και επίσης ε, διακόπτει ο Πρόεδρος και περιμένω την απάντηση στα πολωνικά. Ολοκληρώνει η κυρία Χούμπνερ. Τζίνκουε και μέχρι εκεί φτάνω στα πολωνικά, λέει ο κύριος τζινκουε και μεχρι εκει φτανω στα πολωνικα λεει ο κυριος σιμριμας Θα πρέπει να σας ομολογήσω ότι πολύ λυπάμαι που δεν μιλάω πολεμικά Θα έπρεπε γιατί είμαι γιος ε, ανθρώπου που απελευθερώθηκε από Πολωνούς πριν από 70 χρόνια στην Πρεντά. Αλλά για να απαντήσω ακριβώς ε, στην ερώτησή σας, αυτό που σκοπεύω να κάνω είναι το εξής. Οι ιδέες που έχω για την καλύτερη νομοθεσία θα πρέπει να ξεκινήσει με ένα διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε βήματα για την καλύτερη νομοθεσία. Για παράδειγμα, την μελέτη αντικτύπου που προετοιμάζει. Αυτό θα είναι πάρα πολύ ωφέλιμο για τη δημιουργία ενό νέου συστήματος και θα πρέπει να στραφούμε και προ το Συμβούλιο, αλλά θεωρώ ότι δυστυχώς θα χρειαστεί πολύ πειθό για να μας ακολουθήσει το Συμβούλιο και να ακολουθήσει την ίδια προσέγγιση. Και αυτό είναι απαραίτητο ουσιώδες, γιατί σε αυτή τη φάση προετοιμάζουμε την νομοθεσία και την ελέγχουμε από τον προτέρων, αλλά από τη στιγμή που η νομοθεσία αυτή περάσει από μια μοναδική διαδικασία, νομίζω ότι πουθενά άλλο στον κόσμο δεν υπάρχουν δύο αναγνώσεις, δύο συνομοθέτες, το Συμβούλιο έχει μέλη στη εκτελεστική εξουσία που πηγαίνουν στι Βρυξέλλε. και εν πάση περιπτώσει το σύστημα είναι μοναδικό και περιλαμβάνει διάφορα α, στοιχεία. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και σε εθνικό επίπεδο. Αλλά υπάρχουν αμφιβολίε για τον τρόπο με τον οποίο δρούμε για τη μελέτη εντεκτύπου, για τη σύνθεση της, των ομάδων εμπειρογνωμόνων, για τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Για όλα αυτά λοιπόν υπάρχουν αμφιβολίε και θέλω να είμαι εταίρο του Κοινοβουλίου για τη δημιουργία ενό πιο καλού συστήματο. Αν το παλιό σύστημα είναι παροχημένο, εγώ σίγουρα θα προτείνω να προχωρήσουμε. Αν μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένες αλλαγές με συνεργασία με το Κοινοβούλιο, πολύ καλά. Αλλά ας ξεκινήσουμε το διάλογο και το συντομότερο δυνατόν ας ε, προσπαθήσουμε να περάσουμε τις επιθυμίες ε, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Κυρία Μπρέσο. Ε, Κύριε υποψήφιε αντιπρόεδρε, έχετε ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο και έχετε πει ότι αναλαμβάνετε την υποχρέωση να προχωρήσετε στον τομέα της καλύτερης νομοθεσίας. Πώς θα προσπαθήσετε να μην αγνοήσετε τα βασικά θέματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα. Ε, θα πρέπει να αναζητήσουμε την πλήρη δυνατότητα εκμετάλλευσης των συνθήκων ως έχουν σήμερα και μόνο μεσοπρόθεσμα να μιλήσουμε για την αναθεώρησή τους. Αυτή η στάση είναι κάτι που σας βρίσκει σύμφωνο. Και σχετικά τώρα βλέπετε την επανεξέταση της κατάστασης αυτής στην πρώτη περίοδο της εντολής σας ή στη δεύτερη, ο κύριος Έχω πολλές ερωτήσεις μπροστά μου. Ξεκινώντας νομίζω ότι δεν έχουμε ακόμα χρησιμοποιήσει το πλήρες δυναμικό της συνθήκης της Λισαβόνας. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμα για να πετύχουμε αυτά τα οποία επιθυμούμε. Όταν θα είμαστε σίγουροι ότι δεν μπορούμε πια να κάνουμε τίποτα διαφορετικό, τότε θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μία συζήτηση για την αλλαγή της συνθήκης. Δεν θέλω να προχωρήσω περισσότερο εδώ. Εγώ ενθυμούμαι τις δυσκολίες τις οποίες είχαμε στο παρελθόν. Νομίζω λοιπόν ότι είχα και εγώ προσωπική εμπειρία με τους πολίτες μου για να τους πείσω για το απαραίτητο αυτής της προσπάθειας μετά το 2005 και ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση τότε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό που προσφέρει η ισχύουσα συνθήκη που δεν έχει ακόμα χρησιμοποιηθεί. Σχετικά τώρα με το λεγόμενο fiscal compact λέει, ενώ μιλεί Ιταλικά στα Αγγλικά ο υποψήφιος αντιπρόεδρος. Νομίζω ότι δεν υπάρχει δυσκολία να το εντάξουμε στις ευρωπαϊκές συνθήκες δεν νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη για να υπάρξει, να υπάρξει αλλαγή στις συνθήκες για να το πετύχουμε αυτό. Ο κύριος Κίρκοπ. Κύριε Τίμερμαν, στην ε, mission statement, στη δήλωση της αποστολή σας, είπατε ότι κάθε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα διασφαλίσετε ότι θα σεβέτε την αρχή της επικουρικότητας και αναλογικότητας, καθώς και το χάρτη θεμελιδών δικαιωμάτων. Ως επίτροπος για την καλύτερη νομοθεσία μπορείτε να διασφαλίσετε ότι και κάθε πρόταση θα συνάδει και με την κοινή λογική, γιατί η κοινή λογική στην τελική ανάλυση και η ισορροπία είναι απαραίτητα στοιχεία για να υπάρχει σωστή ε, απάντηση σε πολλωμένου τομεί, όπω για παράδειγμα η μετανάστευση, η ασφάλεια, η δικαιοσία. Τι συγκεκριμένε λοιπόν πρωτοβουλίε σκοπεύετε να λάβετε για να ανακτήσετε την ισορροπία και την εμπιστοσύνη στου Ευρωπαίους πολίτε σε ό,τι αφορά την Ευρώπη και να είναι σίγουροι ότι δεν υπάρχει μόνο δικαιώματα για τα προσωπικά δεδομένα, αλλά και ε, καταπολεμούνται ε, βασικά προβλήματα ότι τηρείται η ασφάλεια δικαιοσύνη των εθνικών συστημάτων και μην, ε, μην ενοχληθείτε να απαντήσετε με την δική μου προφορά του Yorkshire. Έχετε το λόγο. Ο κύριος Τίμερμαντς δεν πρόκειται να αποπειραθώ καν. Η χώρα που γνωρίζετε καλύτερα από όλες είναι και το λίκνο της κοινή λογικής και μετά Πρέπει να πω όμω ότι ακολουθώντα τι πολιτικέ συζητήσει που διεξάγονται στη χώρα σα, αναρωτιέμαι κατά πόσον υπάρχει επαφή με την κοινή λογική. Θα επανέλθουμε σίγουρα σε αυτό το θέμα. Ξέρετε, είμαι πολύ πραγματιστής. Δεν θέλω να είμαι ιδεολόγος για τέτοια θέματα, αλλά θίξατε ένα πάρα πολύ θεμελιώδες ζήτημα, το οποίο θα αποτελέσει και ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα, τα οποία θα κληθούν ε, τα, το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τα επόμενα χρόνια. Οι κοινωνίες μας βρίσκονται υπό άμεση απειλή από άτομα τα οποία συχνά γεννήθηκαν στις κοινωνίες μας και θέλουν να καταστρέψουν τις ε, αξίες μας που δεν θέλουν για παράδειγμα οι γυναίκες να έχουν ίσα δικαιώματα, που δεν τους αρέσει το πώς ε, ε, εγγυόμαστε τα ίσα δικαιώματα για την κοινότητα των ΛΟΑΔ που δεν αρέσκονται στο κράτος δικαίου. Θα πρέπει λοιπόν να προστατέψουμε τις κοινωνίες μας κατά της εξωτερικής αυτής απειλής. Και αν το κάνουμε αυτό θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα πρέπει να θίξουμε τα ίδια τα δικά μας θεμελιώδη δικαιώματα στην πορεία. Αλλά θεωρώ ότι είναι αφελές να πιστεύουμε ότι η ασφάλεια μπορεί να επιτευχθεί μόνο παρατηρώντας και τηρώντας τα θεμελιώδη δικαιώματα. Μπορούμε να προστατεύουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και εκ παραλλήλου να παρέχουμε αυτό που κάθε κυβέρνηση καλείται να παρέχει στους πολίτες της ασφάλεια. Και πιστεύω ότι χρειάζεται να διεξαγάγουμε διάλογο με τα κράτη-μέλη για το πώς θα προσεγγίσουμε το θέμα αυτό, προκειμένου και να τηρούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και να αισθάνονται ασφαλείς στο δρόμο, στα σχολεία οι πολίτες μας. Ευχαριστώ κύριε Σκαβανά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σας δώσω μια νέα ευκαιρία να μιλήσετε τη γλώσσα του Μολιέρου όπως ο κύριος Λάμπερτς. Η ολοκλήρωση της Ευρώπης είναι κάτι σαν τον έρωτα. Χρειάζονται αποδείξεις. Εδώ έχουμε μια χώρα, την Ουγγαρία, η οποία τρεις φορές παραβίασε τις συνδεευρωπαϊκές συνθήκες ελευθερία του τύπου. Έκλεισε μάλιστα πρόσφατα και ένα τηλεοπτικό σταθμό που λέγεται RTL Club γιατί δεν άρεσαν τα σχόλια στην κυβέρνηση. Έκανε έρευνες παράνομες σε ε, μικρές ε, ανθρωπιστικές οργανώσεις της Ουγγαρίας γιατί είχαν πάρει λέει βοήθεια από την Ορβηγία, λες και θα εισέβαλε η Νορβηγία στην Ουγγαρία. Ε, και ταυτόχρονα φορολογία ιδιαίτερη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δεν είναι ουγγρικές και σύν της άλλης μια μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος ε, της Ουγγαρίας με απαράδεκτο τρόπο που καταστρέφει την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος. Έχουμε να κάνουμε με μια συστημική επίθεση στον ευρωπαϊκό κανόνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, ποιο θα είναι ο τρόπος που θα δράσετε, το άρθρο 7 ή κάποιες άλλες διοικητικές δράσεις. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Η ερώτηση αυτή έχει τεθεί τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την Ουγγαρία. Δεν το κρύβουμε αυτό. Είδαμε ότι οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεισέφεραν στο να επιληθούν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα με διάλογο με την Ουγγαρία. Σας διαβεβαίω ότι για την Ουγγαρία όπως και για όλα τα άλλα κράτη-μέλη θα προσπαθήσω να εμπλακώ, να συζητήσω, να συνδιαλλαγώ και να βρούμε τελικά συγκεκριμένες λύσεις για συγκεκριμένα προβλήματα ε, σε στενό διάλογο με το κράτος μέλος. Και δεν θα ε, διστάσω να χρησιμοποιήσω επίσης όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσω την πλήρη και ολοκληρωμένη εφαρμογή και σεβασμό των συνθήκων είναι κάτι ε, το οποίο έχουν προσυπογράψει όλα τα κράτη που είναι μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα παλάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την πλήρη, την απόλυτη τήρηση των υποχρεώσεων που προέρχονται από την προσυπογραφή των κοινοτικών κειμένων από τις χώρες. Κάθε Ευρωπαίος πολίτης έχει δικαίωμα στην απόλυτη εφαρμογή και σεβασμό των δικαιωμάτων του στο σύνολο των κρατών μελών, για όλους τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες. Ο κύριος Χρυσόγονος. Πρόεδρε, η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη με σειρά αποφάσεών της έκρινε ότι μέτρα λιτότητας που επέβαλε στην Ελλάδα η Τρόικα παραβιάζουν κοινωνικά δικαιώματα κατοχυρωμένα στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη αλλά με παρόμοια διατύπωση και στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης οι αποφάσεις αυτές δεν εκτελούνται και μάλιστα η Τρόικα ζητά ολοένα και σκληρότερα μέτρα λιτότητας. Σε σχετική μου ερώτηση, ο Επίτροπος Κατάινεν απάντησε ότι τα έγγραφα του ελληνικού προγράμματος δεν αποτελούν δίκαιο της Ένωσης, υπονοώντας έτσι ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν ισχύουν σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό. Σας ρωτάω λοιπόν, αν κατά τη γνώμη σας η Επιτροπή όταν ενεργεί ως μέλος της Τρόικα δεσμεύεται από το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και αν σκοπεύετε να προχωρήσετε σε ενέργειες για να συμμορφωθεί η Ελλάδα προς τις αποφάσεις της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Uh, Κατά πρώτον, επιτρέψτε μου να πω ότι αν ε, εξετάσετε την κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα, είναι πραγματικά σχεδόν θαύμα το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να ξεπεράσει τις χειρότερες δυσκολίες της κρίσης. Και από ό,τι φαίνεται ότι αυτά που συμφωνήθηκαν μεταξύ της Ελλάδας και της Τρόικας είχαν θετικό αντίκτυπο στην κατάσταση της, Ευρωπα... της ελληνικής οικονομίας δεν ε, κρύβω το γεγονός ότι αυτό είχε μεγάλο τίμημα, βαρύ τίμημα για πολλούς Έλληνες που έχασαν τη δουλειά τους, τα σπίτια τους, τις διεκτησίες τους σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά και πολλοί ακόμα στην Ελλάδα υποφέρουν. Το σχέδιο όμως που ανέπτυξε η Τρόικα, τηρώντας ε, απόλυτα και συμφωνώντας με την, Ευρωπαϊ... με την ελληνική κυβέρνηση, βασίζεται στις συνθήκες και στην κοινωτική νομοθεσία και στις εθνικές ευθύνες της Ελλάδας και πιστεύω, όπως είπε και ο πρόεδρος Γιούγκερ, ότι θα καταστεί, θα είναι απαραίτητο στο μέλλον να ληφθούν περαιτέρω μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρχει καλύτερη και λεπτομερέστατη ανάπτυξη ανάλυση των, του κοινωνικού αντικτύπου των μέτρων αυτών. Αυτό είναι απολύτως ε, κρίσιμο. Αλλά δεν θα έφτανα να πω ότι η Τρόικα ή η Ελλάδα παραβίασαν θεμελιώδη δικαιώματα επιβάλλοντας και συμφωνώντας για ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων για την Ελλάδα. Τούτου λεχθέντος να πω ξεκάθαρα το εξής. Ο χάρτης είναι κάτι το οποίο έχουν προσυπογράψει όλα τα κρατημέλη και ισχύει σε όλα τα κρατημέλη και για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τίμερμανς ε, αναφέρθηκε προηγουμένως ότι η ευρωπαϊκή ευημερία θα πρέπει κατά κύριο λόγο να βασίζεται στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γνωρίζουμε όμως ότι ορισμένα εξ αυτών ε, ξεχνιούνται πολλοί παραμελούν, όπως συμβαίνει πολύ συχνά και με το δικαίωμα σε μη διακριτική μεταχείριση και επίσης και στην ενεργό χρήση της μητρικής γλώσσας. Ένας από τους πολύτιμους θησαυρού Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η πολυγλωσία. Ένας θησαυρό που δεν τον διαφυλάσσουν επαρκώς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ε, μόλις ε, τελείωσε η θητεία μου της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ε, όπου εγκρίναμε ένα μανιφέστο για τα γλωσσικά δικαιώματα που ε, έχει μεταφραστεί αυτό σε 70 γλώσσες. Γνωρίζετε ότι τα γλωσσικά δικαιώματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και εξίσου συχνά παραβιάζονται. Ερωτώ λοιπόν τι προτίθεστε να κάνετε για να προστατεύσετε τα θεμελιώδη δικαιώματα όχι μόνο συγκεκριμένων ε, κρατών αλλά γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτίθεστε να ονοματίσετε τα κράτη-μέλη τα οποία παραβιάζουν αυτά τα δικαιώματα Εντάξει, την καταλάβαμε την ερώτηση, λέει ο πρόεδρος. Ε, παρακαλώ, ο κύριος Τίμερμανς. Κοιτάξτε, ακριβώς όπως και εσείς, ε, και εγώ ε, εκτιμώ ιδιαίτερα την πολυγλωσία, τις πολλές γλώσσες και είχα την τύχη να μεγαλώσω σε μία σειρά ευρωπαϊκών κρατών. Γι' αυτό λοιπόν είχα και την ευκαιρία να μάθω μία σειρά ευρωπαϊκών γλωσσών. Αυτό είναι πραγματικά ένας ανεκτήμητος θησαυρό. Και θα ήταν πολύ λυπηρό εάν μετά από 20-30 χρόνια να, να μιλάμε όλοι μας κακά αγγλικά. Ας μην το κάνουμε αυτό. Ας διαφυλάξουμε τις μητρικές μας γλώσσες και ας προσπαθήσουμε να μιλάμε σωστά αγγλικά και να διδάξουμε τα παιδιά μας να ομιλούν και αυτά γλώσσες όσο καλύτερα μπορούν. Γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχουν προβλήματα με τις γλώσσες των μειονοτήτων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός αυτής. Εγώ έχω συνεργαστεί με αυτά που ήδη έχουμε στα χέρια μας για να προστατεύσω τις γλώσσες των μειονοτήτων και πού μπορούμε με βάση νομικά έγγραφα να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει σεβασμός για γλώσσες μειονοτήτων. Αναφέρομαι στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αναφέρομαι στην, στον ύπατο εκπρόσωπο του ΟΑΣΕ, αναφέρομαι σε ένα Ινστιτούτο Φλέγκσπουργκ νομίζω ονομάζεται, το οποίο με ρημνά για τι μειονότητε. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά εργαλεία. Υπάρχει και ένα, ένας χάρτης ε, του Συμβουλίου τη Ευρώπη, δεν ξέρω αν λέγεται χάρτη, υπάρχει ω κάτι στο Συμβουλίο τη Ευρώπη που ασχολείται με τι γλώσσε των μειονοτήτων. Και αν θέλετε, εγώ ε, θέλω να συνεργαστώ μαζί σα για αυτά τα θέματα, γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά το πόσο στενά συνδέεται η γλώσσα που μιλάει ένας άνθρωπος με την ταυτότητά του και με τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται σε μια κοινότητα. Τώρα, σε μια άλλη γλώσσα μειονότητας, ο κύριος Χέλμερ. Διαρωτώ με κατά πόσον Γνωρίζετε την ε, αγανάκτηση που υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε πάρα πολλού εγκληματίες, του οποίου δυστυχώς δεν μπορούμε να εκδώσουμε. Ε, πολλές φορές επικαλούνται το δικαίωμα τη οικογένειακή ζωής. Όμως και αυτό πια το έχουν τραβήξει όσο δεν πάει άλλο. Υπάρχει ένα Τζαμαικανό 50 ετών, ο οποίο έχει κάνει πολλά παιδιά με διάφορες διαφορετικές γυναίκες ε, και παρόλα αυτά λέει ότι δεν μπορούν να τον εκδώσουν γιατί έχει δικαίωμα στην οικογενική ζωή. Αυτή λοιπόν η κατάσταση οδήγησε στο να υπάρξει δυσφήμιση του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Και θα ήθελα να γνωρίζω εσείς τι δράσεις ε, προτίθεστε να αναλάβετε όταν ε, θα επιβεβαιωθείτε στη θέση σας για να λύσετε κάπως το πρόβλημα και για να διαβεβαιώσετε τους Βρετανούς ότι όσοι απειλούν την κοινωνία μας θα μπορούν στο μέλλον μέλλον να εκδίδονται στη χώρα προέλευσής τους. Ο κύριος Τίμερμανς, κοιτάξτε, αν ε, δούμε λιγάκι την έμπνευση που είχε εκείνος που ε, συνέστησε το Συμβούλιο της Ευρώπης ή κάποιος άλλος που συνέστησε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Είναι το ίδιο άτομο. Νομίζω οφείλουμε πάρα πολλά στον Winston Churchill. Εκείνος είχε την ιδέα ότι θα πρέπει να υπάρχουν και δικαιώματα πάνω από την έννοια του κράτους δικαιώματα που άπτονται άμεσα στους πολίτες ενός κράτους. Αυτό είναι ένα ανεκτήμητο εργαλείο. Ανεκτήμητο για να δοθούν και αποδοθούν δικαιώματα ε, στους πολίτες στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν βέβαια αρνητικά στοιχεία και πρέπει αυτά να τα συζητήσουμε. Γιατί η Βρετανική κυβέρνηση και όταν άλλε κυβερνήσεις λένε ότι βλέπουν να υπάρχουν κάποια αρνητικά στοιχεία και θέλουμε αυτά να συζητηθούν, εμείς το καταλαβαίνουμε αυτό και πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις. Όμως, επιτρέψτε μου να πω και με απόλυτη σαφήνεια, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι ακριβώς επιθυμούμε. Γιατί εάν αφαιρέσουμε την υπεροχή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τότε για τις χώρες όπου δεν τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι χώρες αυτές θα έχουν μια πρόφαση στη συζήτηση, αν θέλετε, ε, που θα γίνει στον Ηνωμένο Βασίλειο, να πούνε, κοιτάξτε, και εμείς δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει αυτά τα δικαιώματα να ισχύουν για τους δικούς μας πολίτες. Άρα δηλαδή φέρουμε ευθύνη απέναντι στο σύνολο των πολιτών στον ευρωπαϊκό χώρο, στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκτός αυτής, έτσι ώστε αυτά που κάνουμε σε εθνικό εθνικό επίπεδο να μην επηρεάζουν τις δυνατότητες πολιτών να έχουν πρόσβαση σε ανθρώπινα δικαιώματα γιατί σε κάποιες χώρες όπως η Ρωσία ας πούμε δεν είναι τόσο αυτονόητο και η Ρωσία δουλεύει, συνεργάζεται με το Δικαστήριο ανθρωπιών Δικαιωμάτων και με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Υπάρχουν κάποιοι χώροι όπου ε, είναι αποδεκτό το κράτος δικαίου. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Σωστά ε, επισημάνεται κάποιες ατέλειες του συστήματος ε, ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κύριος Ντεγκράφ. Κύριε Τίμερμαντς, στις 14 Σεπτεμβρίου ε, μία επιστολή είπατε ότι το Ισλαμικό κράτος ε, δεν έχει να κάνει τίποτα με το Ισλάμ, αλλά παράλληλα οι ευρωπαϊκές, οι ολλανδικές μυστικές ε, υπηρεσίες προειδοποίησαν ότι όσοι πηγαίνουν στη Συρία για να πολεμήσουν έχουν μοναδική ιδεολογία το Ισλάμ. Πού είναι λοιπόν η πηγή του στον Ινδουισμό, στον Χριστιανισμό, αρνείστε τέτοια πιστώσεις της Ολλανδικής Μυστικής Υπηρεσίας και ότι η ροή των μεταναστών με Ισλαμικό ε, υπόβαθρο είναι ενδεχόμενοι τσιχαντιστές. Χτες στη Γερμανία ε, υπήρξαν συγκρούσεις μεταξύ μουσουλμάνων Ισλαμιστών και τσιχαντιστών. Πιστεύετε ότι αυτό δεν αποτελεί κίνδυνο για την Ολλανδική την ασφάλεια και τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν ε, γι' αυτό και πώς μπορούμε να προωθήσουμε το έργο του υποψηφίου Επιτρόπου Αβραμόπουλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Στην παρούσα φάση, στο Κομπάνι, στη Συρία, ε, στα τουρκικά σύνορα υπάρχουν συγκρούσεις, δολοφονίες από το Ισλαμικό κράτος. Και αυτοί που δολοφονούνται είναι μουσουλμάνοι, Κούρδοι, μουσουλμάνοι. Είναι πραγματικά αδιανόητο να μιλάμε για το Ισλαμικό κράτος και να το κάνουμε σύμβολο του Ισλαμικού κόσμου. Και αδικούμε έτσι ένα δισεκατομμύριο μουσουλμάνους βάζοντάς τους στο ίδιο καζάνι. Εγώ ως καθολικός δεν μπορώ να είμαι υπεύθυνο για αυτά που έκανε πριν από κάποιους ε, αιώνους ε, η Ισπανική ε, Εξέταση. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος λοιπόν με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον, την πρόκληση τέτοιων οργανώσεων όπως το Ισλαμικό κράτος. Θα πρέπει να ξεκινάμε με βάση τις δικές μας αρχές, οι οποίες βασίζονται στην εβραϊκή χριστιανική μας παράδοση. Προέρχονται σε μεγάλο βαθμό αυτές οι αξίες από τον κόσμο των μουσουλμάνων. Και έτσι είμαστε σύμμαχοι λοιπόν υπό την έννοια αυτή και χρειαζόμαστε μεν τους δεν. Θα πρέπει μαζί να δράσουμε. Δεν θα πρέπει να ξεκινήσουμε και να σκεφτόμαστε με όρους ε, θρησκευτικού πολέμου. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την άμεση πρόκληση για την ασφάλειά μας. Μέσω των ευρωπαϊκών αξιών, σεβασμός της πολυμορφίας, της ε, ανεξιθρησκείας, των δικαιωμάτων, με τις οποίες έχουμε κατακτήσει, τα οποία έχουμε κατακτήσει με πολλούς αιώνας αγώνα. Uh, <clears throat> uh, uh, Έχω δύο ερωτήσει, κύριε Τίμερμανς να σα κάνω. Η πρώτη, αυτό που αναφέρθηκε η διαθεσμική συμφωνία για την καλύτερη νομοθεσία. Θα ξεκινούσατε φέτος ήδη τις διαπραγματεύσεις και όχι του χρόνου όπως αναφέρετε στις γραπτές απαντήσεις σας προκειμένου η θεσμική συμφωνία να ταιριάξει στο περιβάλλον που δημιουργήσε η συνθήκη της Λισαβόνας. Θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι κατεπήγον. Δεύτερη ερώτηση σε ό,τι αφορά τις ε, εφαρμοστικές πράξεις και τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Οι απαντήσεις σας δεν καθησυχάζουν τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου και λήψη κοινών κριτηρίων. Πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εφαρμόσει τα κριτήρια της συνθήκης σε ό,τι αφορά την κατάρτιση νομοθετικών προτάσεων. Επίσης, πότε και ποια συγκεκριμένα μέτρα πέρα από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων σκοπεύετε να λάβετε για να υπάρξει πρόοδος σε ό,τι αφορά τα θέματα εναρμόνισης. Απάντηση για την πρώτη ερώτηση. Ρωτήσατε κατά πόσον θα ήθελα και θα ήμουν διτεθειμένος να ξεκινήσω να μιλάω με το Κοινοβούλιο για τη Διαθεσμική Συμφωνία για την καλύτερη νομοθεσία πιο σύντομα. Ο μοναδικός λόγος για τον οποίο αναφέρθηκα στο επόμενο έτος είναι γιατί ο πρόεδρος Γιούνκερ ανέφερε ότι θα πρέπει να καταγράψουμε την υφιστάμενη νομοθεσία πρωτίστως και πρωταρχικά και αυτό θα αποτελούσε την πρώτη μου προτεραιότητα. Αν υπάρχει επιθυμία όμως στο Κοινοβούλιο να ξεκινήσουμε πιο σύντομα, είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω έτσι. Καταλαβαίνω το κατεπήγον του θέματος. Αν το Κοινοβούλιο θέλει λοιπόν να ξεκινήσουν πιο σύντομα οι σχετικές διαπραγματεύσεις, προφανώς είμαι στη διάθεσή σας για τις πράξεις κατά και τις εφαρμοστικές πράξεις. Βλέπω και το Γιολάινεν και θυμάμαι όταν καταρτήσαμε τη συνθήκη της Λισαβόνας φαίνονταν πάρα πολύ λογικό να υπάρχει αυτή η διάκριση μεταξύ των άνθρωπων 290 και 291. Στο χαρτί φαίνεται πάρα πολύ λογικό, αλλά καταλαβαίνω και την ανησυχία του Κοινοβουλίου ότι η επιλογή ενός από τα δύο μέτρα έχει ε, συνέπειες για το ρόλο που διαδραματίζει το Κοινοβούλιο. Το κατανοώ απόλυτα αυτό. Και αν γίνει η επιλογή αυτή, Υπάρχει πρόβλημα με το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο θέλει το αντίθετο. Είναι σύγκρουση συμφερόντων και είναι λογικό να υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων και στη μέση είναι η Επιτροπή. Πώ μπορεί λοιπόν να το αντιμετωπίσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πιστεύω ακράδαντα αυτό να είναι λογική και αντικειμενική για τα κριτήρια που εφαρμόζει. Το δικαστήριο δεν μα βοήθησε ιδιαίτερω. Μα είπε βρείτε τα μόνοι σα, λίγο πολύ. Χωρί να θέλω να δείξω ασέβεια προ το δικαστήριο. Λίγο πολύ όμω αυτό μα είπε. Ε, αυτό θα πρέπει να κάνουμε, να τα βρούμε μεταξύ μας. Και καταρχάς θα ήθελα να υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια για να καθορίζεται κατά πόσο πρόκειται για πράξη κατεξιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις. Ο κ. Σίλβα Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, επιτρέψτε μου να σας υποβάλω μία ερώτηση. Και σε αυτή την ερώτηση πρόκειται για τις ε, θεσμικές ε, συνέπειες ε, της οικονομικής διακυβέρνησης. Και εδώ αναφέρομαι σε ευρωπαϊκούς, ε, ευρωπαϊκές οικονομικές δομές. Στη γραπτή σας απάντηση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρεται ότι δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν παράλληλοι θεσμοί στην Ευρωζώνη. Και επίσης είπατε ότι θα έπρεπε να αποφύγουμε μία σειρά θεσμών. Και ρωτώ, σωστά σας ερμηνεύω ισχυριζόμενος ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής, η πρόταση του να υπάρχει κοινοβούλιο μόνο για την Ευρωζώνη είναι κάτι που το απορρίπτεται. Ακριβώς αυτό. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Λίγα μόνο δευτερόλεπτα χρειάστηκα, κύριε Πρόεδρε. Αυτή ακριβώς είναι η θέση μου. Πολύ Ο κύριος Ουζατσόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, μιλήσατε για την καλύτερη νομοθετησία. Μπορείτε να μας δώσετε ίσως κάποια παραδείγματα για κείμενα τα οποία θα πρέπει να εξαφανιστούν πια γιατί παρεμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Και η δεύτερη πρωτοβουλία αφορά τη, δεύτερη ερώτηση, συγγνώμη, αφορά την πρωτοβουλία των πολιτών. Αναφερθήκατε σε αυτό συνοπτικά. Υπάρχει μια προσπάθεια που έγινε από την ε, ε, οργάνωση Ουάνοβας με δύο εκατομμύρια υπογραφές και η οποία αφορά την προστασία της ζωής και απερίφθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρέπει να λειτουργεί αυστηρανομικά, ξερανομικά. ξερά νομικά. Πρέπει να σέβεται τις πρωτοβουλίες των πολιτών της Ευρω... στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω να είστε πιο ανοιχτός απέναντι σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Κύριε Τίμερμανς, έχει το λόγο. Ένα, ένα από τα χειρότερα χτυπήματα στην αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια ήταν κάτι το πάρα πολύ ε, μικρό πράγμα. Had a huge impact on the image of the Όλοι λέγαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ανόητη σε σχέση ε, με <clears throat> μικρά πράγματα ε, και νομοθετούσε όλο σε μικρά πράγματα και για σήμαντα πράγματα και όχι για σημαντικούς νόμους και για σημαντικές παρεμβάσεις. Organization in the Parliament and um, uh, in the Commission. Everyone participating in expert. Ε, νομίζω ότι όσοι συμμετέχουν στις ομάδες των εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να έχουν την κοινή λογική όπως είπε ο κ. Σκέκοπ. Θα πρέπει να έχουν, θα έλεγα, ενστικτοδός την αντίδραση να κατανοήσουν ότι δεν μπορεί να είμαστε τόσο παράλογοι. Δεν θέλω τώρα να περάσω σε πιο συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να προτείνω είναι να αλλάξουμε την κουλτούρα, τον τρόπο με τον οποίο προέρχονται κάποιες από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έρχονται για συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τη δουλειά μας και την εικόνα που δίνουμε προς τα έξω. Σχετικά τώρα με την πρωτοβουλία των πολιτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομικά, επίσημα θα έλεγα, είχε δίκιο απέναντι στην πρωτοβουλία αυτή στην οποία αναφέρατε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν σαφώς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και των υποχρεώσεών της. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορούμε να το συζητήσουμε πολιτικά το θέμα και πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει αυτές τις πρωτοβουλίες έτσι ώστε να γίνει μια συζήτηση με αυτούς οι οποίοι κατέθεσαν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία εμπλέκοντας και αυτό εδώ το κοινοβούλιο. Η κυρία Γκρισμπέκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, λέτε ότι είστε πραγματιστής και ο παδός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα απέναντι στο Συμβούλιο. Αναλάβατε την υποχρέωση να χρησιμοποιήσετε πλήρως τα μέσα τα οποία έχετε στη διάθεσή σας και είπατε επίσης ότι και στα πλαίσια της Ουγγαρίας, της Ουγγρικής περίπτωσης, θα χρησιμοποιήσετε όλα τα άρθρα της συνθήκης και όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, θα ήθελα να επαναλάβετε όμως κάτι εδώ, γιατί όταν ήσασταν υπουργό ε, εξωτερικών στη χώρα σας, ήσασταν κατά των κυρώσεων εις βάρος της Ουγγαρίας. Τι έχει γίνει εν τω μεταξύ. Μια δεύτερη ερώτηση. Είπατε επίσης ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να διασφαλιστεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, βγάλει κάποιους κοινούς δείκτες οι οποίοι με συστηματικό τρόπο θα επιτρέψουν σωστά και την εφαρμογή του άρθρου 7, κάποιους δείκτες λειτουργικούς για όλες τις χώρες. Αναλαμβάνετε λοιπόν την υποχρέωση να προχωρήσετε σε αυτού του είδους την δράση. Καταρχάς, έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κράτος μέλος το οποίο να μην έχει κάποια δεδομένα προβλήματα κάπου κάπου με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τα θεμελιώδη διορθώνω δικαιώματα. Ε, και έχουμε ανάγκη, όλες οι χώρες έχουν ανάγκη, κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο της Ευρώπης που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα να βλέπουν το τι γίνεται και να αναφέρουν τα προβλήματα. Όλες οι χώρες. Τώρα για την Ουγγαρία. Σας είπα, είπα μάλλον στον συνάδελφό σας προηγουμένως, ότι νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε με ε, διάλογο, όπως προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιλύσει με συγκεκριμένο τρόπο τα συγκεκριμένα προβλήματα. Και σε δύο περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέφερε να λύσει τα συγκεκριμένα προβλήματα που είχαν ε, τεθεί στην ε, Ουγγαρία. Δεν τέλειωσε η ιστορία εδώ. Σας είχα πει επίσης και το επαναλαμβάνω ότι εγώ θα χρησιμοποιήσω όλα τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας στο βαθμό που μια χώρα μέλος δεν είναι διατεθειμένη να αλλάξει τη στάση την οποία έχει και την ομοθεσία της όταν είναι αντίθετη του ευρωπαϊκού κανόνα. Σχετικά τώρα με τους κοινούς δείκτες για όλα τα κράτη-μέλη. Εγώ θα προτιμούσα να ξεκινήσουμε από αυτό το ετήσιο συνέδριο. Να δω τι γίνεται με τις άλλες οργανώσεις που ασχολούνται με τα θέματα αυτά στην Ευρώπη. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει ένας θα έλεγα τεράστιος όγκος αναλύσεων στοιχείων που δεν είναι πάντα στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το πρώτο βήμα λοιπόν θα ήταν να δούμε το τι ακριβώς υπάρχει ήδη σήμερα. Εάν καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι κάτι τέτοιο είναι ανεπαρκές, τότε θα κάνω προτάσεις. Αλλά πρώτα παρακαλώ να αναλύσουμε το τι έχουμε στη διάθεσή μας και το τι μέσα είναι σε αυτή την περίπτωση χρήσιμα. Πρόεδρε, κύριε Τίμερμαντς, ε, όταν σας έθεσε μία ερώτηση, κυρία Τσίμερμαν, είπατε για την καλύτερη νομοθεσία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι κοινωνικές διαστάσεις. Αυτό είναι θετικό και είμαι ευχαριστημένος με αυτό. Όταν μιλήσαμε για την Ελλάδα, ε, ξεφύγατε το θέμα της φτώχειας και της ανεργίας που επέφερε η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί. Γι' αυτό λοιπόν δύο συγκεκριμένες ε, συμφωνίες να κάνουμε θέλω. Καταρχάς μπορείτε να μας υποσχεθείτε ότι θα κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας. Όχι μόνο τα κράτη-μέλη αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια να γίνουν ε, μέλη του κοινωνικού χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης και κατά δεύτερον σε ό,τι αφορά την επίσκεψη στο ελεκτικό συνέδριο στο Λουξεμβούργο χθε. Οι κοινωνικοί στόχοι του προγράμματος Ευρώπης 2020 για την καταπολέμηση της στόχιας και της ανεργίας θα τεθούν ως συγκεκριμένες προτεραιότητα στην καλύτερη νομοθεσία. Ο κ. Τίμερμαντ. Στην παρούσα φάση αναμένουμε την γνωμοδότηση του, μάλλον την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Τη στιγμή που θα έχουμε λοιπόν την ε, απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, θα περάσουμε, θα προσπαθήσουμε να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μέλο τη συνθήκη. Νομίζω ότι είναι ύψη της σημασία αυτής και θα είναι το πρώτο μου βήμα. Αυτό τι σημαίνει ότι και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα δεσμεύονται από εκείνη τη στιγμή από όλους τους κανόνες της ε, συνθήκης και θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να γίνει αυτό πλέον. Έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Πρέπει να σας ε, ομολογήσω ότι αυτή η ερώτηση δεν με βρίσκει έτοιμο. Δεν μπορώ να προβλέψω την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό την Κοινωνική Συμφωνία, τον Κοινωνικό Χάρτη, σε ό,τι αφορά τους ε, περιορισμούς που έχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε το θέλουμε είτε όχι. Θα ήθελα να σας υποσχεθώ ευχαρίστω ότι εγώ θα το ελέγξω και θα το μελετήσω το συντομότερο δυνατόν και θα αναλύσω σε τι βαθμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να συνδεθεί και να επικυρώσει αυτό τον κοινωνικό χάρτη και το συμβολίο. Θα πρέπει να σας ομολογήσω με πάσα ειλικρίνη ότι δεν γνωρίζω στην παρούσα φάση επαρκώς τις ε, νομικές συνέπειες και σε ό,τι αφορά τους κοινωνικούς στόχους ε, στην Ευρώπη του 2020 ασφαλώς και αποτελούν ε, αναπόσπαστο σημείο της πολιτικής και του πολιτικού προγράμματος της Επιτροπής Juncker και θα τα συζητήσουμε φυσικά αυτά και με το κοινοβούλιο σας. Η κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω στην ερώτηση τη συναδέλφου για τα βασικά και δικαιώματα στην Ουγγαρία. Είπατε ότι θα πρέπει να διεξάγουμε διάλογο. Ο διάλογος ποτέ δεν είναι αρνητικό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξαγάγουν εδώ και χρόνια διάλογο με το Κοινοβούλιο, με την Ουγγαρία, συγγνώμη σε το περασμένο έτος σε έκθεση του το Κοινοβούλιο είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει τριμερής διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινοβουλίου και Ουγγαρίας και είπατε ο, εξ ονόματος της Ολλανδικής Κυβέρνησης ότι αυτό δεν ήταν απαραίτητο γιατί δεν είχε φτάσει η κατάσταση στην Ουγγαρία σε σημείο που θα σκεφτόμασταν κυρώσεις. Πριν από δύο μήνες ο Βίκτορ στην Ουγγαρία είπε ότι θέλει να έχει ένα κράτος μη φιλελεύθερο. Συγκρίθηκε με τη Ρωσία και με την Κίνα. Η ερώτησή μου λοιπόν προς εσάς είναι η εξής. Δεν πιστεύετε πλέον ότι εδώ υπάρχουν απειλές κατά του συστήματος και ότι τώρα λοιπόν θα πρέπει να λάβει δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μία νέα πρόταση, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου. Ο κύριος Τίμερμανς. αν θα έπρεπε να απαντήσω σε όλα τα σχόλια που κάνει ο Βίκτορ Ορμπάν στις πολιτικές του ομιλίες, θα χρειαζόμουν μια ολόκληρη ημέρα. Τι, τι θα πρέπει να κάνουμε όμως συγκεκριμένα, αν κάτι έμαθα από τον πολιτικό μου πατέρα, τον Μαξ Φαντεστούλ, είναι ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε επακριβέστατα τις νομικές διατάξεις, τις συμπεριφορές των θεσμικών οργάνων σε ό,τι αφορά τους πολίτες. Αυτά θα πρέπει να καταγράψουμε. Εκεί θα πρέπει να κοιτάξουμε κατά πόσο υπάρχει αντίφαση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Τη στιγμή που θα αποφασίσετε ότι θα επικυρωθώ ως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγώ προτίθεμαι να ξεκινήσω τη διαδικασία αυτή. Και φυσικά αυτό θα γίνει με, το κρατης, με τα κράτη-μέλη, γιατί το κράτος μέλος ε, της Ουγγαρίας είναι ένα κράτος μέλος και θα πρέπει να διεξάγεται διά, διάλογος. Ως υπουργό Εξωτερικών, μαζί με άλλους τρεις υπουργούς Εξωτερικών, είχαμε λάβει πρωτοβουλία προκειμένου και στο Συμβούλιο να υπάρχει βάση προκειμένου να εξετάζονται και να πολιτικά ως πώς να συζητιούνται παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων στο Συμβούλιο Τέσσερα κράτη μεταξύ των οποίων και η Ολλανδία λοιπόν έλαβαν την πρωτοβουλία αυτή. Αλλά επαναλαμβάνω, η αρχή γίνεται με τον διάλογο. Και δεν θα διστάσω. Αν δεν υπάρξουν τα αποτελέσματα τα επιθυμητά από τον διάλογο, στη συνέχεια να περάσω στην επιβολή μέτρων. Ε, διαδικασία επί παραβάση, μέχρι και τη δυνατότητα που προβλέπει το άρθρο 7 της συνθήκης, αν παραστεί η ανάγκη. Δεν πρόκειται να φοβηθώ. Γιατί αν ένα πράγμα με ενόχλησε τα τελευταία δέκα χρόνια είναι η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δείχνει έντονη πυγμή και να μιλάει πάρα πολλά για κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά πάντα να τηρεί πιο διστακτική στάση σε ό,τι αφορά τη δική μας εσωτερική κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θελήσει να βάλει ένα τέρμα και να κάνει μια αλλαγή με συγκεκριμένα πολιτικά μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Ελμάρα. Κύριε Τίμερμαν, διερωτώ με κατά πόσον θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης προκαλεί μεγάλες ε, αδικίες γιατί ανατρέπει δικαιώματα Βρετανών εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως ε, το δικαίωμα δίκης ε, με ενόρκους. Ε, σε οι δύο, δύο μου πήγαν και στάλησαν σε άλλη περιοχή και κατά την διάρκεια που κρατούντο δεν τους δόθηκε δίκαιη δίκη, ούτε είχαν και διερμηνία, ούτε και λεπτομέρειες για το κόστος που προέκυψε. Έτσι λοιπόν, εγώ ισχυρίζομαι αυτό που σας είπα, ότι τελικά δεν δικαιολογείται η έκδοσή τους. Οι άνθρωποι αυτοί πέστησαν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά και αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα, υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα. Σήμερα οποιοδήποτε Βρετανός ε, μπορεί να εγκλειστεί χωρίς να έχει δικαίωμα έφεσης. Ε, εσείς λοιπόν κύριε Τίμερμαν, τι ακριβώς θα κάνετε για να αναχαιτήσετε αυτή την αδικία. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δεύτερη ερώτησή σας. αν θέλετε αυτό που ρωτήσατε τώρα ήταν ε, ο καθρέφτης αυτού που ρωτήσατε προηγουμένως. Είπατε προηγουμένως ότι η Ευρώπη δίνει πάρα πολλά δικαιώματα στους πολίτες ε, της χώρας σας και τώρα όμω λέτε ότι η Ευρώπη δεν δίνει αρκετά δικαιώματα. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Αν πραγματικά θέλουμε να καταπολεμήσουμε το έγκλημα στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, χρειαζόμαστε επιγόντως το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Και είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε και υγιείς νομικές εγγύησεις ε, διαφύλαξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων για εκείνους που συλλαμβάνονται με βάση ευρωπαϊκό ένταλμα Προφανώς ε, δεν μπορώ να αναφερθώ με λεπτομέρειες ε, στην περίπτωση που αναφέρατε. Όπως το παρουσιάσατε είναι πραγματικά τραγική η περίπτωση αυτή, αλλά ε, και εγώ δεν μπορώ να τοποθετηθώ πάνω σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ισχυρίζομαι όμως ότι επειδή αντιμετωπίζουμε πάρα πολλές απειλές και επειδή το οργανωμένο έγκλημα έχει πολλές δυνατότητες να εξαπλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα, πόσο μάλλον σε ευρωπαϊκή, η καταπολέμηση του εγκλήματος στην Ευρώπη είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη. Και να σα πω την αλήθεια, εγώ το βρίσκω αυτό μία από τι μεγαλύτερε επιτυχίε μα στον τομέα τη καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο. Ο κύριο Λεμπρετόν έχει το λόγο. Κύριε Τίμερμαν, ο πρόεδρο Γιούνκερ είπε ότι είστε το δεξί του χέρι. Γι' αυτό θα είστε ένα υπερεπίτροπο που θα έχει δικαίωμα βέτο, αρνησή κυρία, στι πρωτοβουλίε των συναδέλφων του μη αναμενόμενη η προαγωγή σας. Την πήρατε όμως γιατί κάποιες χώρες όπως η Γαλλία έχουν πάρα πολλούς δισταγμούς σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είστε διπλωμάτης, είστε ευγενής, αλλά όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προεδρεύεται πλέον από τον πρώην διαχειριστή ενός φορολογικού παραδείσου. Είστε μια ευκαιρία λέμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα αποτύχετε κύριε Τίμερμανς γιατί η προσπάθεια αυτή ενημερωτική την οποία κάνετε και διαφημιστική δεν θα κοροϊδέψει κανέναν. Πώς μπορεί να υπάρξει μια πραγματική επικορικότητα όταν θα υπάρξει μια δικτατορία μια ενισχυμένης λιτότητας από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ουσία θα δώσετε περισσότερα δικαιώματα ε, εσείς σε κάποιους ολιγάρχες και σε κάποιες μειονότητες ε, σε σχέση με τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση σε αυτά που είπατε. Ίσως να υπάρχει μια ερώτηση, θα απαντήσω σε αυτό, αν και ίσως αυτό το οποίο θα σας πω θα το κρίνετε ότι είναι άχρηστο. Αλλά για τα επόμενα πέντε χρόνια και εφόσον το Κοινοβούλιο με επιφορτήσει με την συγκεκριμένη αποστολή, Άλλωστε να πω εδώ ότι αν ενθυμούμε καλά, ε, την εποχή των γονιών μου, τα μέλη της οικογένειάς μου, ε, δεν μπορούσαν να κοινωνικοποιηθούν γιατί ήταν γκέι, γιατί είχαν συγκεκριμένο, συγκεκριμένο σεξουαλικό προσανατολισμό. Τους έδερναν στο δρόμο λόγω ακριβώς αυτού του προσανατολισμού τους. Ενώ σήμερα στις περισσότερες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι άνθρωποι του ιδίου φύλου έχουν το δικαίωμα να νυμφεύονται. Είναι κάτι το οποίο για μένα είναι η έκφραση ε, ε, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ξεκάθαρα ευρωπαϊκή αντίληψη θα έλεγα, προέρχεται και από τα αποτελέσματα της Γαλλικής Επανάστασης, βασίζεται ακριβώς σε θεμέλια τα οποία έστησαν χώρες όπως η Γαλλία Ανθρώπινα δικαιώματα για όλους, άνδρες και γυναίκες. Έτσι έλεγε αυτός ο άνθρωπος που ε, δολοφονήθηκε ο Ζων Ζορές ε, εδώ και 100 χρόνια από ανόητους εθνικιστές. Αυτή μας, αυτός μας μίλησε για τις ατομικές ελευθερίες και η Γαλλία αυτή την αντίληψη πρέπει να την έχει και να είναι υπερήφανοι για αυτήν. Χάρη στην Γαλλία βρισκόμαστε εδώ σε αυτό το επίπεδο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Äh, η κυρία Lange. Ναι, ναι, ναι, εξ όσο γνωρίζω είμαι ακόμα γυναίκα, ναι. Η κυρία Lange. Και θα θέσω την ερώτηση στη μητρική μου γλώσσα. Συχνά μου ακούμε ότι οι ακράσεις αυτές ε, είναι αντιεκλειστήντα εσωτερικής πολιτικής. Ε, να πω ότι παρόλο που δεν είμαι από δική σας πολιτική οικογένεια, ελπίζω να τα πάτε πάρα πολύ καλά. Είπατε ότι η Ευρώπη πλήττεται από έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και αυτή η εμπιστοσύνη μπορεί να ανακτηθεί μόνο αποδεικνύεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αξιόπιστη και γι' αυτό λοιπόν καθήκον σας είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικεντρωθεί στα καθήκοντα τα βασικά, ενέργεια, απασχόληση, ανάπτυξη. Αυτά λένε οι πολίτες ότι θα πρέπει να κάνει η Ευρώπη, όχι να κοιτάει τις λεπτομέρειες. Είδαμε λοιπόν ε, την ε, γοητεία σας και την ε, γλωσσομάθειά σας σήμερα και πολλά θα πετύχετε, αλλά θέλω να ξέρω στην τελική ανάλυση, όταν θα υπάρχουν προτάσεις που δεν θα μπορέσετε να περάσετε, θα έχετε τη δύναμη να αντισταθείτε και ποια συγκεκριμένα, σε ποια συγκεκριμένα θέματα μπορώ να σας κρίνω εγώ σε πέντε χρόνια. Mijn eerste opdracht is Πρώτο μου καθήκον είναι ασφαλώς να φροντίσω προκειμένου κάθε επίτροπος να είναι επίτροπος για την καλύτερη νομοθεσία. Γιατί μόνο αν κάθε επίτροπος στο δικό του τομέα αρμοδιότητα λάβει υπόψη ότι θα πρέπει να φροντίσει να είναι καλύτερη η νομοθεσία και πιο αποτελεσματική, πιο αποτελεσματική μόνο τότε θα πετύχουμε. Δεν πρόκειται να λειτουργήσει αυτό αν ε, περιμένετε να κάνουν το σερίφι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να εξαναγκάσουν τους ε, συναδέλφους να κάνουν πράγματα που δεν θέλουν να κάνουν. Θα πρέπει ως σώμα να φροντίσουμε προκειμένου να υπάρχει λιγότερη νομοθεσία όπου δεν είναι απαραίτητη αυτή και να φροντίσουμε η Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα και όχι μόνο ε, φανταζή. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ε, συλλογική διοίκηση στην Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έχει δικαίωμα να καθορίζει την ατζέντα. Το Σώμα των Επιτρόπων έχει δικαίωμα να καθορίζει την ατζέντα τη Επιτροπή και θα πρέπει λοιπόν να καθοριστεί το τι είναι αρκετά όριμο θέμα για να μπει στην ατζέντα και φυσικά θα κοιτάξω ποια μέτρα είναι απαραίτητα και αν είναι απαραίτητα κατά πόσο είναι αυτή η σωστή μορφή πρόταση ε, των ε, μέτρων. Το βέτο ξέρετε είναι κάτι το περίεργο, δεν ε, λειτουργεί αν απειλεί κανεί με αυτό θα πρέπει να υπάρχει, αλλά ποτέ να μην χρησιμοποιείται ως απειλή, ποτέ να μην χρησιμοποιείται γενικά. Ήμουν στην Ολλανδία τμήμα ε, και συμμετείχα σε δύο ε, κυβερνήσεις ε, συμμαχίας. Επισήμως η Ολλανδική κυβέρνηση λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία. Σε δύο λοιπόν κυβερνήσεις συμμαχικές ε, δεν χρειάστηκε ούτε μία φορά να γίνει ψηφοφορία γιατί με τρόπο συλλογικό λαμβάναμε αποφάσεις. Ελπίζω λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τέτοιο τρόπο συλλογικής διαχείρισης να καταφέρουμε να πετύχουμε αυτά που έθεσε ως ε, στόχο και συμφώνησε μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Jean-Claude Juncker στο mission statement του. Okay. Αγαπητέ κύριε Τίμερμαν, στην εισαγωγή σας είπατε ότι αυτές οι ακροάσεις ε, είναι η καλύτερη ώρα της ε, Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Το ίδιο ίσχυσε και για τους υποψήφιους πριν από τις τελευταίες εκλογές. Ε, βεβαίως οι βασικότεροι υποψήφοι αυτοί που έβαλαν υποψηφιότητα για την Προεδρία της Κομισιόν δεν ήρθαν από τα 28 κρατημέλη, αλλά πολύ πιο λίγα. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, ε, πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό εκλογικό δίκαιο και το δεύτερο ερώτημα που θέλω να σας υποβάλω είναι το εξή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πάρα πολλά δικαιώματα, αλλά όχι το δικαίωμα ε, να αναλαμβάνει νομοθετικές πρωτοβουλίες. Αυτό είναι δικαίωμα της Κομισιόν. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ, ε, σε ε, πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε, παραδείγματος χάρη στην πρωτοβουλία για τους πολίτες, είπατε ότι πρέπει να υπάρχει ευρεία συζήτηση. Στις δικές μας τις εκθέσεις απλά γίνεται μία ανακοίνωση και μετά το πράγμα υποτίθεται ξεχνιέται ή καταλήγει κάπου σε κάποιο γραφείο. Τι έχετε να πείτε από αυτού. Ο κύριος Τίμερμανς, κοιτάξτε, όσον αφορά τους υποψήφιους για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, μπορεί κανείς να πει ότι θέλει. Εγώ ήδη συζήτησα από αυτού με τον πρόεδρο. Ένα πράγμα γνωρίζω με σαφήνεια. Χωρίς τους υποψήφιους για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή η Επιτροπή δεν θα ερχόταν ποτέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα πολιτικά του κόμματα ήταν σε θέση να ορίσει ποιος θα γίνει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ ότι υπήρξε μια δημοκρατική ανανέωση και ξέρετε πολύ καλά κύριε Λάινεν τι σημαίνει το προηγούμενο. Όταν υπάρχει προηγούμενο κάτι δεν μπορεί πλέον να ανασταλεί. Παρότι λοιπόν έχω κάποιες αμφιβολίες σχετικά με τις δημοκρατικές συνέπειες των υποψηφίων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρετε, το γεγονός αυτό δεν οδήγησε να πάνε στις εκλογές να συμμετάσχουν περισσότεροι Ευρωπαίοι, όμως παρόλα αυτά εδώ στους ευρωπαϊκούς θεσμούς οι επιρροές ήταν σημαντικές και αυτό είναι καλό. Τώρα, κατά πόσον όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν στο να υπάρξει ευρωπαϊκό εκλογικό δίκαιο, δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί επί του θέματος να αναλάβει πρωτοβουλία. Ίσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά σίγουρα τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που θα μπορούσαν να αναλάβουν την πρωτοβουλία, κάτι που δεν προβλέπεται με συνθήκη. Ως προς το άρθρο 225, ρωτήσατε πώς αντιδράει η Κομισιόν σε προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά εσείς είπατε ότι οι αντιδράσεις ε, πολλές φορές ε, είναι ευσύνοπτες, ε, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Κοιτάξτε, ίσως πρέπει να υπάρχει καλύτερη αντίδραση στις δικές σας τις πρωτοβουλίες. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει, σαν διαδικασία όμως μπορώ να το φανταστώ. Κοιτάξτε κύριε Τίμερμανς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα ε, να καταθέσει προτάσεις. Όσον αφορά τώρα αυτά που είπε ο κύριος Τίμερμανς, νομίζω ότι μπορούμε να επανέλθουμε αργότερα. Ο κύριος Σίπελ ε, εγώ έχω ερωτήσεις ε, και από τους δικούς μου του συναδέλφους. Αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών είναι ένα νέο εργαλείο στο να μπορούν ε, να συμμετέχουν οι πολίτες ε, στη λήψη αποφάσεων. Όμως δυστυχώς αυτό δεν πετυχαίνει. Και εσείς είπατε ότι η Κομισιόν έχει το δικαίωμα να απορρίπτει κάποιες πρωτοβουλίες. Το C34 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί λοιπόν το απέρριψε τι θα κάνετε για να ξεκινήσει η πολιτική συζήτηση που όπως είπατε κι εσείς είναι απαραίτητη. Τι θα κάνετε εσείς προσωπικά για να εξυπηρετήσετε τα δικά μας ε, τα προσωπικά συμφέροντα. Κοιτάξτε, η φύση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών είναι η εξής. Ζητάνε από την Επιτροπή να καταθέσει πρόταση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν εκλήθη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κατέθεσει πρόταση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Άρα δηλαδή καθαρά τυπικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αναγκασμένη να αντιδράσει όπως αντέδρασε στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Μία πρωτοβουλία δεν αποτυγχάνει βέβαια όταν υπάρχει κάποια αντίδραση της Επιτροπής. Η πρωτοβουλία ε, μπορεί να ληφθεί όταν πολλοί άνθρωποι συνενώνται γιατί πιστεύουν ότι κάτι είναι σημαντικό. <clears throat> Η Κομισιόν βέβαια έχει το δικαίωμα τυπικά να πει όχι, παρόλα αυτά ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι Κομισιόν μπορούν να συνεχίσουν τον διάλογο με εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία. Νομίζω λοιπόν αυτή τη δυνατότητα θα πρέπει να την χρησιμοποιούμε περισσότερο στο μέλλον. Και θέλω να επαναλάβω το εξή. Η πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών όσο έχει παγιωθεί στη συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρει ότι η πρωτοβουλία σημαίνει ότι η Κομισιόν καλείται να καταθέσει πρόταση. Αυτό βέβαια πρέπει να βασίζεται πάνω σε ένα νομικό πλαίσιο ε, στο οποίο να μπορεί να λειτουργήσει η Κομισιόν και όλα αυτά ορίζονται από τα σχετικά άρθρα της συνθήκης. Ο κύριος Γκέρενς έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σχετικά με την ε, εξωτερική εκπροσώπηση της ζώνης ε, ευρώ είπατε ότι πολλά κράτη-μέλη δεν είναι ιδιαίτερα διατεθειμένα να εμπλακούν προς την κατεύθυνση αυτή. Πώς σκοπεύετε να ξεπεράσετε τις δυσκολίες αυτές και να ενισχύσετε σε εξωτερικό επίπεδο τη ζώνη ευρώ. Και τέλος σχετικά με την ανεξαρτησία της Σκοτίας. Προς το παρόν αποφεύγετε την απάντηση ε, και δεν συζητάτε για το θέμα της πιθανής απόσχησης περιφερειών από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά στα πλαίσια και του δημοψηφίσματος του Βρετανικού το 2017. Ε, πώς ε, ε, θα πρέπει να πάρετε κάποια μέτρα στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει μια κάποια απόσχηση. Κύριε Τίμερμαντς, έχετε το λόγο. Η εκπροσώπηση, η εξωτερική εκπροσώπηση σε διεθνές επίπεδο, στο διεθνές θέμα, σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό να σας ε, πω ότι αυτό σίγουρα θα πάρει κάποιο χρόνο. Μία σειρά κρατών μελών που έχουν το ευρώ στο νόμισμα τους έχουν δική τους εκπροσώπηση, για παράδειγμα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και σε κάποιες περιπτώσεις ε, στα πλαίσια αυτά υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες είναι εξωτερικές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια. Άρα η αναδιάρθρωση όλου του συστήματος ασφαλώς θα πάρει χρόνο. Αλλά φυσικά μπορούμε να αναρωτηθούμε αν αλλάξει το σύστημα αυτό. Και αν υπάρξει ένας εκπρόσωπος για όλη την Ευρωζώνη, θα μειωθεί έτσι ο αντίκτυπος και η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε πραγματιστές. το πώς ε, θα δράσει η Ευρωζώνη όταν θα ομοδοποιηθούν όλα τα κράτη-μέλη σχεδόν θα ε, έχει σημασία και θα, έχει, θα ανακύψει το ερώτημα αυτό και θεωρώ λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανέλθει στο ύψο των περιστάσεων σε ό,τι αφορά τώρα το δικαίωμα να βγει κανείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση το χειρώθηκε στην συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν είναι φυλακή η Ευρωπαϊκή Ένωση αν ένα κράτος μέλος θεωρείς ότι το συμφέρει καλύτερα να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει το δικαίωμα να το πράξει. Δεν λέω ότι αυτό αποτελεί κάτι το οποίο είναι δικαιολογημένο και ότι πρέπει να συμβεί, αλλά κάθε κρατός μέλος μπορεί να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν είναι... Ε, φυλακή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σπινέλη. Eh, Ευχαριστώ κύριε Τίμερμανς. Επαναλαμβάνω την ερώτηση που έθεσαν ήδη δύο συνάδελφοι ε, από την Ελλάδα μάλιστα γιατί η απάντηση δεν είναι πλήρης. Πράγματι θέλετε χρόνο για την ε, υπογραφή της ε, συνθήκης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Τα δικαιώματα των πολιτών υφίστανται επιθέσεις, ιδιαίτερα τα κοινωνικά. Εκτός και αν πράγματι πιστεύετε ότι η συμφωνία με την Τρόικα και η παρέμβασή της είχε θετική ε, επίπτωση στην Ελλάδα για τα θεμελιώδη δικαιώματα υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε αυτά τα οποία λέτε εσείς ότι υπήρξε σεβασμός των κοινοτικών κανόνων και αυτά που είπε ο Επίτροπος Κατάινεν ότι στην περίπτωση της Τρόικα δεν εφαρμόζονται οι κοινωνικές ρυθμίσεις. Εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι το όνομα Σπινέλη με εμπνέει πάντα. Γνώρισα τον Αλτιέρο Σπινέλη από μικρό παιδί και δεν θα τον ξεχάσω ποτέ. Πρόκειται για μια, πραγματι... για μια πραγματικά εντυπωσιακή προσωπικότητα που οικοδόμησε την Ευρώπη που όλοι ξέρουμε σήμερα. Τώρα για την εφαρμογή, τον, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, μπορεί να γίνει. Έχουμε να κάνουμε με ευρωπαϊκό δίκαιο, με δεδομένες ρυθμίσεις. Στις δράσεις τους ε, οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να σέβονται το κρατούν δίκαιο και που περιλαμβάνονται και στην χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα στην δράση των ευρωπαϊκών οργάνων. Σχετικά με την Ελλάδα τώρα. Είμαι πεπισμένος ότι οι κοινωνικές συνέπειες των μέτρων είναι τρομερές. Η χώρα αυτή υποφέρει, το γνωρίζουμε αυτό, το βλέπουμε αυτό. Ξέρουμε ότι έχουν χάσει τη δουλειά τους, έχουν προβλήματα επιβίωσης και χωρίς την βοήθεια από πλευράς των οικογενειών δεν θα ήταν κάτι τέτοιο εφικτό. Υπάρχει λοιπόν μια συζήτηση που γίνεται, βλέπω ποιες είναι οι κοινωνικές επιπτώσεις αυτών των μεταρρυθμίσεων. Όμως οι μεταρρυθμίσεις αυτές ήσαν απαραίτητες. Δεν έγιναν οι μεταρρυθμίσεις αυτές από την Ελλάδα και την Τρόικα γιατί ήθελαν να χτυπήσουν τον πληθυσμό της Ελλάδας. Έγιναν οι μεταρρυθμίσεις γιατί η Ελλάδα βρισκόταν σε μια οικονομική κατάσταση φρικτή. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι απαραίτητες και βλέπουμε και κάποια θετικά πλέον αποτελέσματα. Πασκάλ Ντυρό. Κύριε Τίμερμανς, η Ευρώπη δεν έχει την αξιοπιστία, δεν, δεν έχει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών έχει πάρα πολλές ε, αδυναμίες ε, και υποκύπτει στα λόμπι εύκολα. Πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και αυτό εξαρτάται από την υποδειγματική συμπεριφορά των ε, ευρωπαϊκών οργάνων. Στη βασική του ομιλία σας επιφορτίζει ο κύριος Γιούνκερ να συντονίσετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εδώ εντάσσεται και το θέμα της συγκρούσεως συμφερόντων. Ο κώδικας συμπεριφοράς απαγορεύει σε επιτρόπους να ασχολούνται με θέματα τα οποία άπτονται ε, των προσωπικών του συμφερόντων και ενασχολήσεων, αλλά δεν καλύπτεται το θέμα των συζύγων, της ή του συζύγου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μπορείτε λοιπόν να τροποποιήσετε αυτόν τον κώδικα καλής συμπεριφοράς, έτσι ώστε να καλύπτονται τα λεγόμενα οικογενειακά οικονομικά συμφέροντα και όχι μόνο τα ατομικά. Και δεύτερον, θέλετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της σύγχρονης δημοκρατίας να είναι ένας χώρος ο οποίος κατέχει τα απαραίτητα στοιχεία έτσι ώστε να μπορεί να κρίνει την οικονομική ανεξαρτησία των επιτόπων. Ο κ. Τίμερμανς απαντά λέγοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει μια ανάλυση των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των ιδίων των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αν δεν κάνω λάθος και είναι μια ανάλυση η οποία νομίζω είναι συγκρίσιμη με αυτήν την οποία κάνουμε εμεί στο εσωτερικό της Επιτροπής. Σχετικά με τη διαφάνεια τώρα. Και εγώ θέλω να αυξηθεί η διαφάνεια. Αλλά αυτό θα πρέπει να το πετύχουμε από κοινό. Ας προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τις πρακτικές στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως και στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Και τότε θα δούμε ποιο είναι το όργανο το οποίο είναι σε καλύτερη θέση για να πει στους άλλους ότι πρέπει να κάνει ένα βήμα περισσότερο. Νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής να προχωρήσουν από κοινού δεν πρέπει να υπάρχει καμία παρανόηση σχετικά με την προσωπική αξιοπρέπεια των μελών του Κοινοβουλίου και των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν μπορέσουμε να το κάνουμε με τον καλύτερο κοινό δυνατό τρόπο, γιατί όχι να το συζητήσουμε για να το πετύχουμε. Αλλά σε επίπεδο νομικό το να πούμε εμείς ποια είναι η οικογένεια και πού φτάνει το οικογενειακό συμφέρον Ξέρετε ότι από χώρα σε χώρα υπάρχουν τεράστιες διαφορές στα πλαίσια αυτών των ορισμών. Το τι θεωρεί κανείς οικογένεια δηλαδή νομικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να οριστεί, το κατανοείτε αυτό. Παρ' όλα αυτά θέλω να είμαι συνεργάτη σας και εταίρος σας, έτσι ώστε να αποδείξουμε προς τα έξω ότι τα δύο όργανα θέλουν να υπάρξει η πληρέστερη δυνατή διαφάνεια έτσι ώστε να πείσουμε το Συμβούλιο, το οποίο έχει πάρα πολλή δουλειά να κάνει, θα έλεγα, να κάνει αυτά τα οποία εμείς έχουμε κάνει και εσείς έχετε κάνει. Μπορέλη. Και εγώ πρέπει να σας πω δεν μπόρεσα να μην ενδώσω στον πειρασμό να σας κάνω και μία δεύτερη ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσοντας τις δραστηριότητες της ε, ε, έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες. Ε, βεβαίως, θέλω να πω ότι εδώ πρόκειται για πράξεις οι οποίες έχουν πολύ σημαντικές συνέπειες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Η Επιτροπή λοιπόν πώς προτίθεται να βεβαιώνει και να διαφυλάσει ότι όλες αυτές οι πράξεις θα διαφυλάσσονται ε, με έναν πολύ επικοδομητικό τρόπο. Κοιτάξτε, πρέπει να κάνω μία ανάλυση τι γίνεται με αυτές τις πράξεις. Γιατί γνωρίζω ότι πάρα πολλές πράξεις είναι πολύ τεχνικές. Δεν έχουν ε, πολιτικές ή οικονομικές ε, προεκτάσεις. Είναι όμως απαραίτητες οι πράξεις αυτές για τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως εκεί όπου οι πράξεις αυτές ε, ασκούν επιρροή, όπως ισχυριστήκατε κι εσείς, ε, επηρεάζουν τους επιχειρηματίες, τους πολίτες, εκεί πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι πράξεις αυτές ελέγχονται με δημοκρατικό τρόπο είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Άρα δηλαδή εγώ ε, θέλω να κάνω την ανάλυση όλων αυτών των πράξεων για να διαπιστώσω ποιες είναι αυτές οι πράξεις που έχουν προεκτάσεις και απαιτούν τη δημοκρατική επαλήθευση είτε από το Ευρωπαϊκό είτε από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτό θα αποτελεί ένα τμήμα της δουλειάς μου να βρούμε μια διαθεσμική, διοργανική μάλλον συμφωνία για καλύτερη νομοθεσία. Better regulation. Ο κύριος Σοπφλίν. Η κυβέρνηση της Ολλανδίας ε, έχει ήδη ε, δηλώσει ότι δεν θα υπάρχει πια Ευρώπη σε 54 περιοχές. Και εγώ διερωτώ με ποια είναι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε εθνικές και ευρωπαϊκές ε, ενωσιακές αρμοδιότητες. Πώς μπορούμε να βρούμε μια ικανοποιητική λύση και για τις δύο πλευρές ε, και αυτό κατ' ουσία είναι και το βασικό πρόβλημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε λιγάκι τον τρόπο με τον οποίο νομοθετούμε. Επίσης, πρέπει στην αξιολόγηση των επιπτώσεων της νομοθεσίας μας να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Γιατί αν μπορέσουμε να φέρουμε σε φως τις επιπτώσεις ε, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή σε πολίτες. Αν δηλαδή το γνωρίζουμε αυτό έγκαιρα, τότε αυτό θα βοηθήσει πολύ στο να αποφασίζουμε κατά πόσον θα προχωρήσουμε με μια συγκεκριμένη νομοθεσία ή όχι. Επίσης πιστεύω ότι η αξιολόγηση των επιπτώσεων είναι αναπόσπαστο τμήμα όλου του νομοθετικού έργου. Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προτείνει άλογο και στο τέλος της διαδικασίας να προκύψει ε, Καμίλα. Γιατί, διότι παρεμβαίνει το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σίγουροι ότι παραγγέλνουμε άλογο και προσφέρουμε στους πολίτες άλογο και όχι καμήλα. Η ενδιάμεση λοιπόν αξιολόγηση είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει στη συζήτηση να συμμετέχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Δεν είμαι σίγουρος ότι οι ομάδες συμφερόντων που μιλάμε εδώ στις Βρυξέλλες, ότι αυτές οι ομάδες εκπροσωπούν πάντα ε, τα συμφέροντα των κρατών μελών. Νομίζω ότι υπάρχει ε, ένα είδος ε, θεσμοθετημένου λόμπι στις Βρυξέλλες και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό να καταγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι εκπρόσωποι ομάδων ποιησης ε, που βρίσκονται στις Βρυξέλλες και αυτό να είναι γνωστό οποτεδήποτε προετοιμάζεται ε, μια νομοθετική πράξη. Αυτό λοιπόν αφορά τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Μωράες έχει το λόγο. Κύριε Τίμερμανς, νομίζω ότι η απάντησή σας αποκάλυψε κάτι για τη στάση σας ε, ε, προασπίζεστε τις αξίες μα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά θα ήθελα να πάω λίγο παραπέρα και να σα ρωτήσω το εξή. Σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και την προάσπιση του τι είδου επίτροπο θα είσαστε όταν υπάρχει η απειλή του Ισλαμικού κράτου, ότι υπάρχουν και άλλα ε, βασικά προβλήματα και δεν ε, μιλάμε μόνο για τους ε, νόμους στην Ουγγαρία που δεν μεταφέρονται για τη λιτότητα, τα δικαιώματα των σεξουαλικών μειονοτήτων, των ΛΟΑΔ. Τι σκοπεύετε να κάνετε για τα θέματα αυτά. Θα είσαστε επίτροπος, αντιπρόεδρος που θα υπερασπιστεί αυτές τις θεμελιώδεις αξίες. Θα είσαστε το άτομο αυτό που θα υπερασπιστεί το, τις θέσεις μας σε δύσκολους καιρούς ε, λιτότητας. Εμείς οι Ευρωπαίοι μπλέκουμε η απάντηση. Σε όλη μας την ιστορία μπλέκαμε. Ψάχνουμε κάποιον να κατηγορήσουμε κάθε φορά. Είναι κομμάτι της ανθρώπινης φύσης, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Και υπάρχει τόση πολυμορφία στην Ευρώπη που πάντα θα βρούμε κάποιον να κατηγορούμε. Τους Εβραίους, τους Μουσουλμάνους, τους Χριστιανούς, τους Γκέι, τις γυναίκες τους ε, Ρώμα, τους ε, ΣΥΝΤΙ, πάντα κάποιον βρίσκουμε να κατηγορήσουμε. Ο θρίαμβος της, ε, του ευρωπαϊκού πολιτισμού είναι ακριβώς να περιορίσει αυτή την αντίδραση και να δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο εντός του οποίου μπορούμε να ελέγξουμε αυτή την εγγενώς ανθρώπινη αντίδραση. Καθώς μάθαμε ότι δεν είναι σωστό να σκοτώνουμε. Μάθαμε ότι και καλό είναι να μην μεταχειριζόμαστε διακριτικά τους ανθρώπους. Αλλά αυτό συνεχώς ανακύπτει σε περίοδους κρίσεων και πάντα κάποιον άλλον βρίσκουμε να κατηγορήσουμε για τα προβλήματά μας. Η Ευρώπη λοιπόν αυτό ακριβώς έχει ως σκοπό να καταπολεμήσει αυτή την αντίδραση. Αν αυτό με καταστήσει μη δημοφιλή, ε, τι να κάνουμε. Αλλά αν δεν προασπίσει τον θεμελιώδη δικαιώματα σήμερα, δεν πρόκειται να υπάρχει αύριο Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί επί της ουσίας είμαστε μια ένωση αξιών και το γεγονός ότι τα τελευταία 30-40 χρόνια έχουμε προσεγγίσει ε, και ιδιαίτερα μετά την πτώση του τείχους του Μπαρολίνου, αυτό έχει γίνει κυρίως σε ό,τι αφορά τις κοινέ μας αξίες. Αν είχα πει πριν στους παππούδες μου πριν από 30 χρόνια ότι στην αλλαγή του ε, επόμενου αιώνα στην Ολλανδία θα μπορούσαν να παντρευτούν άτομα του ίδιου φίλου, θα με βάζανε στο τρολοκομείο. Και τώρα αν πω στα παιδιά μου, όταν μιλάω στα παιδιά μου, δεν μπορούν να φανταστούν ότι στην Ολλανδία δεν θα ήταν δυνατόν αν αγαπιούνται δύο άντρε να μπορούν να παντρευτούν. Έτσι έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Καλό είναι αυτό και αυτό θα πρέπει να προστατεύεται δια νόμου. Σας ευχαριστώ κύριε Τιμπερμάνς και κύριε Μάκινταϊρ. Κύριε Τιμπερμάνς, εδώ είμαι. Από αυτά που μας είπατε σήμερα, νομίζω ότι και εσείς είστε επεπισμένος όπως και εγώ ότι μπορούμε να αναπτύξουμε πολύ περαιτέρω το δυναμικό της Ευρώπης αν απαλλάξουμε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από το περιττό κόστος και τη γραφειοκρατία που που επιβάλλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο. Το Κοινοβούλιο ε, ενέκρινε έκταση της Επιτροπής Απασχόλησης που έκανε διάφορες συστάσεις για ένα πιο φιλικό περιβάλλον για δημιουργία θέσεων απασχόλησης για να υπάρξει πιο πολλή δράση, για να περιοριστεί η γραφειοκρατία και επίσης εγκρίναμε ψήφισμα για τις ε, δέκα... Διαδικασία διαβούλευση και είπαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να θέσει στόχους για να μειωθεί μέχρι το 2020 κατά 30% η γραφειοκρατία. Αυτό το υποστήριξαν πολλέ οργανώσει επιχειρήσεων, CBI, Συμμαχία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. δεδομένη λοιπόν τη ευρεία αυτή της θα δεσμευτείτε για να μπει ένα στόχο για να περιοριστεί το ρυθμιστικό βάρος της επιχειρήσης στο επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Τίμερμαντς. Όπως σας είπα, θα είμαι οτιδήποτε λειτουργεί θα το υποστηρίξω και αν υπάρχει δυναμικό να πετύχουμε αποτελέσματα θα το υποστηρίξω. Εδώ πέρα όμως να βάλω και να σας επισημάνω και το εξή. Σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδιαίτερως, δεν νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ενθουσιώδης σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα ως τώρα των δράσεών μας. Να δούμε λοιπόν τι έχουμε κάνει έως τώρα. Γιατί από τότε που ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ μου ζήτησε να αναλάβω τα καθήκοντα εφόσον με επιβεβαιώσετε στο ρόλο μου αυτό, εξετάζω την κατάσταση και τόσος κόσμος μας λέει ότι μα έχουμε κάνει τόσο πολλά πράγματα και τελικά όταν μιλάω με τις επιχειρήσεις είναι εντελώς διαφορετικό. Εντελώς διαφορετική εντύπωση που προσλαμβάνω. Άρα θα ήθελα συγκεκριμένα μέτρα για, για να απαλλαχθούν από το φόρτο τους οι επιχειρήσεις, προκειμένου ο χασάπης, ο φούρναρης να αισθανθούν λιγότερο βάρος. Κάτι άλλο να προσθέσω. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ειλικρινία και στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό, γιατί πολύ εύκολο είναι να κατηγορούμε την ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το βάρος αυτό, το φορτίο αυτό. Πόσο συχνά όμως αναγκάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση γιατί το ζητούν τα κράτη-μέλη. Γιατί θεωρούμε ότι η πρόταση αυτή προέρχεται από ομάδες συμφερόντων και τελικά δηλώνουν αυτές οι ομάδες συμφερόντων ότι δεν τις χρειάζονται την νομοθεσία αυτή. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε με μεγάλη προσοχή το θέμα της επαφής μας με τα άτομα αυτά που προσπαθούμε να βοηθήσουμε. κυρία Βίξτρομ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές ήσαν, θα έλεγα, ένα ξυπνητήρι για όλους μας. Πρέπει να ακούσουμε επιτέλους τους πολίτες της Ευρώπης. Σαν πρόεδρος της Αρμόδιας Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να πω ότι η Επιτροπή μου σε καθημερινή βάση ε, έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλές αναφορές ε, από το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε σχέση με την εφαρμογή και τον σεβασμό του κοινοτικού νόμου. Έχουμε να κάνουμε με ένα χρυσορυχείο στοιχείων δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να βελτιωθούν οι νομικές ρυθμίσεις που ισχύουν. Είστε υπεύθυνοι λοιπόν για την καλύτερη νομοθεσία στην Ευρώπη. Δύο ερωτήσεις. Πρώτον, πώς θα βελτιώσετε τη συνεργασία ανάμεσα στα δύο θεσμικά μας όργανα, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε με καλύτερο τρόπο την Επιτροπή Αναφορών και δεύτερον, τι σημαίνει για σας προσωπικά η έννοια της καλύτερης νομοθετικής δραστηριότητας. Για την πρώτη σας ερώτηση, αν με καλέσετε στην Επιτροπή σας θα έρθω. Αν θέλετε να μελετήσω τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις τις οποίες ε, είχατε μέχρι τώρα θα το κάνω. Αν θέλετε γενικά εγώ να κάνω ε, ένα σχόλιο για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργήσουν ε, οι αναφορές θα το κάνω, όχι σε ατομική βάση βέβαια, γιατί οι συγκεκριμένες αναφορές ε, έχουν κάποιους νομικούς περιορισμούς και δεν είμαι σε θέση να τους σχολιάσω δημόσια. Αλλά αν υπάρχουν κάποιες γενικές τάσεις τις οποίες βλέπετε, αυτό θα με βοηθήσει, θέλω να τις ξέρω. Θέλω να γνωρίζουμε πού υπάρχουν προβλήματα έτσι ακριβώς να πάρουμε τα μέτρα τα οποία είναι χρήσιμα. Ίσως η Επιτροπή πρέπει να κατηγορηθεί, ίσως κάποιο, άλλη, κάποιο άλλο επίπεδο. Συνήθως βέβαια στρέφονται οι κριτικές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν με προσκαλέσετε λοιπόν θα είμαι εταίρος σας σε αυτή την προσπάθεια. Τώρα το τι σημαίνει για μένα καλύτερη νομοθεσία. Αυτό το οποίο σημαίνει ότι κάποιος που είναι φούρναρης, να μην χάνει μισή ολόκληρη μέρα για να συμπληρώνει έγγραφα και να κάνει το ίδιο για τρία διαφορετικά όργανα και υπηρεσίες και να μπορεί να διαχειρίζεται τον φούρνο του με σωστό τρόπο και να προσλαμβάνει και νέους εργαζομένους. Ευχαριστώ. Τσβίφκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα σύντομα να επανέλθω στην νομοθετική διαδικασία στην οποία αναφερθήκατε στην πρώτη σας ομιλία και στις δράσεις τις οποίες θα πρέπει να αναλάβουμε από κοινού έτσι ώστε να απλοποιήσουμε το νομικό σύστημα. Παράλληλα με αυτό θα πρέπει να σεβαστούμε και την αρχ... τις κάποιες αρχές όπως η αλληλεγγύη, η αναλογικότητα οι κοινωνικές πολιτικές ε, ε, και η πολιτική περιβάλλοντος. Και αυτό είναι απαραίτητο να το κάνουμε για να μην έχουμε υπερβολική γραφειοκρατία και να μην ξεπεράσουμε τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προβλέπετε λοιπόν να δημιουργήσετε ένα ανεξάρτητο, ανεξάρτητο σύστημα παρακολούθησης ε, της εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων και νόμων ένα όργανο ανεξάρτητο δηλαδή, εκτός Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί όταν είναι κανείς απ' έξω βλέπει καλύτερα. Και ο Στίμερμανς. Η αλληλεγγύη πράγματι σημαίνει τα πάντα για όλους. Νομίζω ότι το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε το τι ακριβώς σημαίνει η επικουρικότητα. Νομίζω ότι μπορούμε να υποφεληθούμε ε, από τη στενή επικοινωνία με τα κοινοβούλια των κρατών μελών όπου η ε, αναλογικότητα και η επικορικότητα ελέγχονται συστηματικά. Υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης. Πιστεύω ότι οι μεμονωμένοι επίτροποι θα πρέπει να πηγαίνουν στα κοινοβούλια των κρατών μελών αν έχουν σηκώσει κάρτες κίτρινες ή κόκκινες ή πορτοκαλί μάλλον θα πρέπει να παίρνουν πληροφορίες, να ενημερώνονται ε, και οι ενημερώσεις αυτές να είναι χρήσιμες και για μας την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αναλύουμε συγκεκριμένα το ποιος είναι ο ρόλος της επικουρικότητας. Αυτός είναι ο στόχος και της νέας διοργανικής συμφωνίας για την καλύτερη νομοθετική λήψη νομοθετικών αποφάσεων το αν είναι απαραίτητο να υπάρξει μια ανεξάρτητη υπηρεσία που να ελέγχει τη σωστή εφαρμογή. Δεν νομίζω να είμαι ειλικρινής. Αυτό το οποίο όμως νομίζω είναι ότι απαιτείται μεγαλύτερη διαδραστικότητα ανάμεσα στα κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, εγώ ήμουν έξι φορές βουλευτής στην Εθνική Βουλή των Κάτων Χωρών. Στην αρχή το σύστημα δεν υπήρχε, ενώ σήμερα είναι αρκετά περίπλοκο και επιτρέπει να ελέγχεται ο βαθμός σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας και της αρχής της αναλογικότητας. Είναι κάτι όμως το οποίο δεν θα πρέπει να γίνεται και αντικείμενο κατάχρησης αν κάποιοι δεν ε, δέχονται κάποιες από τις προτάσεις που γίνονται. Η ε, επικουρικότητα και ο έλεγχος της επικουρικότητας αφορά όχι το αν μια πρόταση είναι καλή ή κακή, αλλά για το αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρμόδια ή όχι. Τσίπελ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσίμερμαν. Καλωσορίζω σήμερα την ε, δεσμευσή σας ε, ε, σχετικά με τη διοργανική συμφωνία απέναντι στο Συμβούλιο της Ευρώπης και την Επιτροπή της Βενετίας. Όμως, ίσως μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για τα εξής. Τι θα κάνετε για να διασφαλίσετε ότι ο μηχανισμός κράτος δικαίου θα είναι ένας μηχανισμός ε, για διαχείριση κρίσεων με σωστές παρεμβάσεις, ένας ε, μηχανισμός που θα προβλέπει καλύτερες ε, δυνατότητες κυρώσεων στην περίπτωση που διαπιστώνεται συστηματική παραβίαση των αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και στην περίπτωση που αποτυγχάνουν τα συστήματα ελέγχου και ισορροπιών στα κράτη-μέλη. Πώς μπορείτε λοιπόν να διασφαλίσετε ότι ένας τέτοιος μηχανισμός θα ισχύσει όλα τα κράτη-μέλη με ίσους όρους και με διαφάνεια. κύριε Στιμεμάνης, κοιτάξτε, είναι σαφές νομίζω ότι αν δρώντας ή ολιγορώντας, αν η Κομισιόν ε, προκαλεί την εντύπωση ότι επιλέγει κάποια κράτη-μέλη και αγνοεί άλλα, αυτό θα σημαίνει ότι το σύστημα έχει αποτύχει. Πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και ακριβείς ε, στον τρόπο που κρίνουμε και όχι διότι ε, κάποια κρατημέλη ε, προκαλούν πολύ ε, να τους βάλουμε στο μάτι ή επειδή κάποια άλλα είναι πολύ μεγάλα για να τα αμφισβητήσει κανείς. Στην περίπτωση αυτή, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αυτό ε, θα υπονομεύσει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να είμαστε σχολαστικοί στην αμεροληψία μας, ακριβείς στις αναλύσεις μας και να βασιζόμαστε σε πολύ συγκεκριμένε νομικές διατάξεις και προδιαγραφές. Μπορούμε να υποφεληθούμε από τη δουλειά άλλων οργανισμών και όπως σας είπα, γίνεται πολύ καλή δουλειά από διάφορους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και από ΜΚΟ, από τον ε, Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και άλλους. Σε τελική ανάλυση υπάρχουν τα εργαλεία. Υπάρχει δυνατότητα να επιβάλλονται κυρώσεις. Υπάρχει η δυνατότητα να καταφύγει κανείς στο άρθρο 7 αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι νέες διαδικασίες, πολιτική βούληση χρειαζόμαστε για να εφαρμόζονται αυτά που ήδη υπάρχουν. Και ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα δοκιμαστούμε κατά τα επόμενα έτη για να αποδείξουμε κατά πόσον έχουμε την πολιτική αντοχή, κατά πόσον μπορούμε να ζητάμε από τα κράτη-μέλη να ανταποκρίνονται σε αυτά που έχουν υπογράψει. Ε, διότι εάν έχει κανείς υπογράψει και επικυρώσει μία συνθήκη προφανώς και είναι υπόλογος. Η κυρία Κοράτσα. Σας ευχαριστούμε πολύ που δείξατε ότι θέλετε να αλλάξετε λιγάκι το σύστημα, ε, πράγματι είναι απαραίτητο να είμαστε αποτελεσματικοί και να υπάρχει και εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ερωτώ λοιπόν συγκεκριμένα, ποια είναι τα προγράμματά σας για να διασφαλίσετε ότι τα κράτη-μέλη θα εφαρμόζουν τις οδηγίες και δεν προσθέτουν απλά περισσότερη γραφειοκρατία. Θα είναι αυτό ε, προτεραιότητα για σας. Επίσης αυτή η φοβερή θέση που τα έχετε θα σημαίνει ε, μεγαλύτερη ιεράρχηση ή θα σημαίνει ότι ε, θα επιβάλλεται στα κρατημέλη να εφαρμόζουν τους κανόνες. Πρόσβαση στα έγγραφα, ε, μη διακριτική μεταχείριση με βάση την, ε, τις πολλές αρμοδιότητες, άραγε τα οριζόντια δικαιώματα πραγματικά θα ε, παρισφρήσουν στην κουλτούρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά όλα αυτά, ο τρόπος που ρωτήσετε μου θυμίζουν μία πρώην συνάδελφο από τη που δεν θα αποκαλύψω βέβαια το όνομά της. Κοιτάξτε, αν θέλουμε να είμαστε επιτυχείς πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Θα ήθελα να είμαστε ιδιαίτερα διαφανείς στον τρόπο με τον οποίο νομοθετούμε. Θέλω να υπάρξει διοργανική συμφωνία με το Κοινοβούλιο για να διασφαλίσουμε ότι θα εφαρμόζουμε την αρχή της ενδελεχούς εξέτασης των προτάσεών μας. Και θέλω να υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θέλω οι μικρές επιχειρήσεις να πούν για δες κάτι λειτουργεί. Έχει περιοριστεί το διοικητικό άκτος, γιατί όσο δεν λέγεται αυτό, ό,τι και να κάνουμε δεν θα είναι τόσο επιτυχημένο. Όσον αφορά τώρα την ε, προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, γνωρίζετε ότι ε, αυτό είναι ένα αναπόσπαστο στοιχείο ε, στις αρμοδιότητες όλων των επιτροπών. Εγώ θα έχω μια οριζόντια, θα έχω οριζόντιες αρμοδιότητες, θα μπορώ δηλαδή να πω τους επιτρόπους να βλέπω κατά πόσον λαμβάνουν υπόψη τους τα θεμελιώδη δικαιώματα και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι όλα αυτά θα ενταχθούν ε, στην καθημερινότητα των επιτρόπων. Ε, συζητήσαμε μεταξύ μας για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών, παραδείγματο χάρη, οριζόντιο θέμα και αυτό. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν βελτιωθούμε στο να διασφαλίσουμε την προστασία των παιδιών μας τα επόμενα χρόνια, αν δεν επιδείξουμε συγκεκριμένα στοιχεία με ποιο τρόπο προστατεύουμε τα παιδιά που είναι πολύ ευάλωτα στην κοινωνία, οφείλουμε να το κάνουμε αυτό, γιατί με τον τρόπο αυτό ε, θα υπηρετήσουμε καλύτερα ε, τους ε, νέους στην κοινωνία μας. Η κυρία Φαγιόν. Σας ευχαριστώ κύριε Τιμερμάν. Θα ήθελα να περάσουμε στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της μετανάστευση. Προτείνατε για να διασφαλίσετε ότι όλοι οι μετανάστες που καταφτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να είναι να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα ανεξάρτητα από το φύλλο, τη κοινωνική τους προέλευση, την ε, πεποίθηση, τη θρησκεία, σεξουαλικό προσανατολισμό, αναπηρία κτλ. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών πώς θα χρησιμοποιήσετε τις αρμοδιότητά σας για να αντιμετωπίσετε το θέμα της διακριτικής μεταχείρισης ε, κάποιων ε, ομάδων στην κοινωνία μας, ιδιαίτερος των Ρωμά. Η απάντηση θα ήθελα να πω και να ξεκινήσω από το δεύτερο ερώτημα που θέσατε. Πριν από χρόνια, όταν εργαζόμουν για τον ΟΑΣΕ για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, γράψαμε μια έκθεση για την ε, κατάσταση των Ρωμά και των Σύντη ευρωπαϊκή, στον ευρωπαϊκό χώρο. Ήταν πραγματικά ντροπιαστικά τα αποτελέσματα. Συνδυασμός φρικτών διακριτικών μεταχειρήσεων ε, κοινωνικού αποκλεισμού, αυτοαποκλεισμού σε κάποιες περιπτώσεις από την ε, εκπαίδευση και από άλλους τομείς της ε, κοινωνίας. Αυτά πριν από 20 χρόνια. Κοιτώντας τι γίνεται σήμερα. Νομίζω ότι πολλά, πολύ λίγα έχουν αλλάξει για τους Ρωμά και τους Σύντη στην Ευρώπη και νομίζω ότι όλη η Ευρώπη είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Αποτύχαμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση με φρικτό τρόπο, συλλογική ευθύνη. Μια και δεν μπορούμε να του θεωρήσουμε πολίτες μίας συγκεκριμένης χώρας μόνο. Με, σε συνεργασία με, άλλες, ε, με άλλα ευρωπαϊκά όργανα προτίθαμε να δω πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση για τους Ρωμά και του Συντη. Σήμερα λοιπόν που μιλάμε για κατάχρηση κοινωνικών συστημάτων και αυτούς τους οποίους κατηγορούμε συχνά και στους οποίους επιβάλλουμε σκληρά μέτρα είναι συχνά οι Ρωμά που δεν έχουν πολλές ε, φορές που να πάνε. Και σε ό,τι αφορά τους Ρωμά έχουμε λοιπόν τεράστιο έργο ακόμα να κάνουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όλοι έχουν, τα ίσα, έχουν δικαιώματα σε ό,τι αφορά την προστασία των θεμελιωτών δικαιωμάτων. Αλλά να πούμε ότι υπάρχει, και να είμαστε ειλικρινεί γι' αυτό, ότι υπάρχει μεγάλος πειρασμός ε, για την παρανομία. Η παρανομία ενδεχομένως να είναι μια κερδοφόρος κατάσταση για κάποιες ομάδες στις κοινωνίες, αλλά αυτή η παρανομία ε, καθιστά αδύνατο να εφαρμοστούν από πλευρά της κοινωνίας και των ε, οργάνων της κοινωνίας τα θέματα προστασίας και θα πρέπει να είμαστε και πιο δραστηροί σε ό,τι αφορά επιχειρηματίε που προσλαμβάνουν παράνομα άτομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο ε, Ράγκελ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Τίμερμαν, διάβασα τα άρθρα σα, τι ανακοινώσει σα, την ομιλία σα. Εσείς ε, βλέπετε ποιες είναι οι απόψεις των εταίρων σας για το θέμα της επικουρικότητας και για τις εξουσίες ε, του Κοινοβουλίου. Η αρχή της επικουρικότητας επειδή συνδέεται με το βέλτιστο επίπεδο αποδοτικότητας δεν έχει σαν στόχο τον περιορισμό των δράσεων της Ένωσης αλλά την διεύρυνση των δραστηριοτήτων της. Το ξεχνάτε αυτό ε, πάρα πολύ συχνά φοβάμαι. Η επικουρικότητα, εφόσον γίνει σωστή κατανοητά, σημαίνει περισσότερες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα θέτω το ερώτημά μου. Τι συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύετε να αναλάβετε έτσι ώστε να ενισχύσετε τον ρόλο των κοινοβουλίων των κρατών μελών και ποια μέλη προβλέπετε έτσι ώστε ο κομβικός ρόλος των ε, κοινοβουλίων δεν θα υπονομεύσει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχάς οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι εγγεγραμμένες θα έλεγα βαθιά μέσα στη συνθήκη, δεν μπορεί να αμφισβητηθούν. Υπάρχει μια κάποια τάση ιδιαίτερα και από το όργανο το οποίο καμιά φορά εγώ εκπροσωπούσα, να κάνουμε προτάσεις οι οποίες φαίνονται καλές αλλά δεν είναι πολλές φορές απαραίτητες. Εγώ θέλω αντίθετα τώρα πια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει προτάσεις στους τομείς που θεωρούνται κατά προτεραιότητα σημαντικοί και να γίνεται αυτό το οποίο είναι απαραίτητο να γίνει. Ίσως έχω διαφορετική αντίληψη για την επικουρικότητα από ότι εσείς. Έχουμε διαφορετικές απόψεις για την ίδια βασική αρχή. Παρ' αυτά υπάρχουν τομείς όπως η πολιτική ενέργειες που είναι εγγεγραμμένες και αυτές αγκυρωμένες στη συνθήκη. Οπότε ε, απαιτείται ευρωπαϊκή δράση εκεί. Η βασική μου αντίληψη για την επικουρικότητα είναι ότι μπορεί κανείς να αναλάβει η δράση σε υψηλότερο επίπεδο εφόσον το υψηλότερο αυτό επίπεδο είναι το μοναδικό το οποίο ε, θα ε, δώσει ε, αποτελέσματα. Και μπορεί σε ευρωπαϊκό κανείς επίπεδο να βρει μια λύση που δεν μπορεί να βρει σε εθνικό επίπεδο. Τώρα, για τη δεύτερη ερώτησή σας, και ίσως εδώ να σας αδικήσω λίγο γιατί δεν κατανόησα πολύ καλά αυτό που είπατε. Νομίζω, ε, θυμάμαι τις συζητήσεις που γινόντουσαν στην αρχή της συνέλευσης για την Ευρώπη, για τη συνθήκη και για τους ανταγωνισμούς Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα τελευταία χρόνια η αίσθηση που έχω είναι ότι υπάρχει μια σαφέστατη εταιρική σχέση και συνεχώς βελτιούμενη ανάμεσα στα κοινοβούλια και το ευρωπαϊκό και πρέπει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Και όπως είπα ή προσπάθησα να πω στις εισαγωγικέ μου παρατηρήσεις, η Ευρωπαϊκή αυτή Ένωση δεν θα οικοδομηθεί εις βάρος και εναντίον της βούλησης των κρατών μελών και των πολιτών. Ε, πρέπει να εμπλακούμε λοιπόν με τα κοινοβούλια διότι είναι οι εταίροι μας και θα μας βοηθήσουν να κάνουμε αυτό που θέλουν οι πολίτες. Ρέγνα. Μία ερώτηση για το Ρεφίτ κύριε Τίμερμαν. Στην ανακοίνωσή της για το ρεφίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται και σε κάποιες συμφωνίες επίσης για τους κομμωτές, σαν παράδειγμα, ε, στα πλαίσια της καλύτερης νομοθετικής ρύθμισης, γιατί η συμφωνία αυτή θεωρείται ε, εμπόδιο για την επιχειρηματικότητα αλλά δυστυχώς αυτό είναι κάτι το οποίο ε, σαν ε, πρόταση θα δημιουργήσει προβλήματα σε επίπεδο δικαιωμάτων εργασιακών και συνθήκων εργασίας και υγείας κτλ. Πρέπει οι καλύτερες λοιπόν ρυθμίσεις να δίνουν τα δικαιώματα που θα οδηγήσουν με τη σειρά τους σε ένα ασφαλή ε, χώρο εργασίας και τι σκοπεύετε να κάνετε για να μειώσετε το διοικητικό βάρος που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες χωρίς να επηρεάσετε αρνητικά τα κοινωνικά στάνταρτς για τους υπαλλήλους και τους καταναλωτές. Το καλύτερο δεν θα πρέπει να σημαίνει συστηματικά λιγότερο ή και τίποτα, ιδιαίτερα όταν διακυβεύονται κοινωνικά επίπεδα προστασίας και περιβάλλοντος. Σα ευχαριστώ για τι παρατηρήσει σα. Πράγματι η καλύτερη νομοθεσία δεν είναι μη νομοθεσία και δεν πρέπει να υπάρχει ει βάρο τη κοινωνική προστασία και τη προστασία του περιβάλλοντο. Αυτό το είπα πολλέ φορέ. Καταλήγεται όμω σε κάποια συμπεράσματα σε σχέση με την πρωτοβουλία για του κομμωτέ, όπω την λέμε. Νομίζω ότι ήταν μια ιδέα η οποία δημιουργήθηκε στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη ζητήθηκε να κάνει μια πρόταση, αλλά τα κράτη-μέλη είναι σε θέση ή δεν είναι σε θέση να διασφαλίσουν την προστασία στον χώρο εργασίας των κομωτών. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή μήπω είναι ένα επιπλέον παράδειγμα όπου οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν λύσεις σε εθνικό επίπεδο και προσφεύγουν στην Ευρώπη για να κάνουν κάτι. Δεν είμαι λοιπόν βέβαιος ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να συνεχίσουμε. Νομίζω ότι υπάρχει πολιτικός χώρος για τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δώσουν μια απάντηση θετική. Εφόσον το επιθυμούν βέβαια. Εάν πιθανώς εγώ στο μέλλον γίνω επίτροπος θα πρέπει να διασφαλίσω ότι η δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι μια ανταπόκριση ευρωπαϊκή απαραίτητη. Είναι χρήσιμο για την Ευρώπη να κάνει κάτι τέτοιο ή γιατί δεν τα κάνουν τα κράτη-μέλη αυτό. Υπάρχει εσωτερική αγορά για τους κομμωτές που απαιτεί ευρωπαϊκές δράσεις είναι κάτι το οποίο πρέπει να οργανώσουμε σε αυστηρά εθνικό επίπεδο και αν τεθεί το ερώτημα και καταλήξει η πλειοψηφία στο ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα το σταματήσω εγώ αυτό, πρέπει να είμαι πρακτικός και να το κατανοήσω. Όμως η πολλαπλότητα των αντιλήψεων, των πολιτισμών και των πρακτικών σε μία πρώτη φάση θα με κάνει να σκεφτώ ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να το αντιμετωπίσουν αυτό σαν θέμα. Ευχαριστώ κύριε Τίμερμαν, ο κύριο Γιάρ. Εδώ είμαι. Για το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων με βάση το άρθρο 51 θα πρέπει να εφαρμόζεται το κοινοτικό δίκαιο και ο χάρτης ε, θεμελιωδών οικημάτων έγινε δεσμευτικός με την συνθήκη της Λισαβόνας. Και έτσι λοιπόν έρχονται όλο και περισσότερες αναφορές στο Κοινοβούλιο που αναφέρονται σε αυτό το χάρτη. Όμως ένας μεγάλος αριθμός των αναφορών ε, δεν καλύπτει τα κριτήρια του άρθρου 51, απορρίπτονται οι αναφορές και δεν μπορεί να γίνει τίποτα και στα κράτη-μέλη. Πολλοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι το άρθρο 51 είναι ασαφές, νεφελώδες ναι, και αισθάνονται ότι περιορίζεται τα δικαιώμα, δικαιώματά τους αναφορά. Εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό? Και πώς μπορεί κανείς να εξηγήσει στους Ευρωπαίους πολίτες ότι το δικαίωμα του αναφέρεστε, ε, που το έχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει πλέον όρια με βάση των, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και κάτι άλλο, ε, μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένας ανεξάρτητος οργανισμός ο οποίος να ασχολείται με την αξιολόγηση, με τον έλεγχο ε, της αξιολόγησης των επιπτώσεων και λυπάμαι αυτά που αστέλωσε ήταν και με σαξονική διάλεκτο, όχι γερμανικά. Κοιτάξτε, όσον αφορά τις ε, αναφορές, θα ήθελα να συνεργαστώ με την πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να δω πού υπάρχουν τα προβλήματα με το άρθρο 51. Όμως ότι υπάρχουν ε, κάποια όρια στο δικαίωμα το αναφέρεστε, αυτό υπάρχει και σε εθνικό επίπεδο και στα κράτη-μέλη γίνεται κάτι τέτοιο. Κατά πόσον είναι σαφές το δικαίωμα όχι, αυτό δεν μπορώ να το αξιολογήσω. Όμως ε, αν υπάρχουν δυσκολίες με το άρθρο 51, ευχαρίστως να το συζητήσουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Όταν καλούμεθα να αξιολογήσουμε κατά πόσον μία πρόταση θα οδηγήσει εκεί που επιθυμούμε, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αποφαίνεται επαγγελματικά και αμερόληπτα. Να υπάρχει και απόσταση από κάποια συμφέροντα και να υπάρχει και τεχνογνωσία. Όλα αυτά πάντα αφορούν την Κομισιόν. Ε, τεχνογνωσία, απόσταση από συμφέροντα, αμεροληψία και όταν υπάρχει μια τέτοια αξιολόγηση και ε, έχει αντιδράσει η Κομισιόν, θα ήθελα και εγώ ε, αυτά να τα μοιράζομαι με το Κοινοβούλιο, να τοποθετήσετε κι εσείς, να μας λέτε κατά πόσο λειτουργήσαμε σωστά ή όχι. Και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αυξήσουμε τη διαφάνεια. Ευχαριστούμε κύριε Τίμερμαντς, η κυρία Δελβό. Κύριε Τίμερμαντς, είμαι εξ αριστερών. Να επανέλθω στο θέμα της επικουρικότητας. Σας ευχαριστώ που διευκρινίσατε ακριβώς την άποψή σας και ότι θέλετε να διευκρινιστεί ακόμα περισσότερο η έννοια της επικουρικότητας και στη γραφτή σας απάντηση είπατε ότι θέλετε να βελτιώσετε τη διαδραστικότητα με τα, ευρωπαϊκά, με τα εθνικά κοινοβούλια. Εμείς είμαστε υπέρ φυσικά της ενίσχυσης του ρόλου των κοινοβουλίων των κρατών μελών για να έρθει η κοινοτική πολιτική κοντά στους πολίτες. Και γιατί θέλουμε να προχωρήσουμε ε, στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ο φόβος μου είναι αντίθετος από τον προηγούμενο τι θα κάνετε έτσι ώστε ο σεβασμός της αρχής της επικουρικότητας να μην χρησιμοποιηθεί σαν άλοθη για να καθυστερήσουν οι εξελίξεις που θα οδηγήσουν στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Τίμερμαντς. Κοιτάξτε, ο κίνδυνος είναι προφανής. Είναι προφανής ο κίνδυνος στα διάφορα κράτη-μέλη, σας το είπα αυτό. Είπα ότι γνωρίζω συγκεκριμένες περιπτώσεις, ακόμα και στις χώρες που γνωρίζω καλύτερα, όπου χρησιμοποιείται η επιχειρηματολογία που λέγει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αρμόδια στο συγκεκριμένο τομέα. Ακριβώς όμως το κάνουν αυτό γιατί δεν τους αρέσει η ουσία της πρότασης. Είναι μια καταχρηστική θα έλεγα παρουσίαση των αρμοδιοτήτων των κοινοβουλίων και με βάση την αρχή της επικουρικότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρμόδια για να κάνει τέτοιου είδους προτάσεις και φυσικά πρέπει να βασιζόμαστε στη συνθήκη για να τις κάνουμε τις προτάσεις αυτές. Υπάρχει και η αναλογικότητα εδώ. Η, το μέσο το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να το πετύχουμε αυτό είναι το κατάλληλο για να πετύχουμε τον στόχο τον οποίο έχουμε θέσει. Αυτά είναι νομίζω τα στοιχεία της ανάλυσης η οποία γίνεται από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα πρέπει να διευκρινιστεί αυτό το πράγμα μαζί με τα κοινοβούλια των κρατών μελών, γιατί πολλές φορές χρησιμοποιείται το θέμα σαν άλοθη για να απορριφθούν οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ο έλεγχος επί της ουσίας και το δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μαζί με το Κοινοβούλιο να νομοθετεί και της Επιτροπής να κάνει προτάσεις νομοθετικές δεν θα πρέπει να απεισχναθεί από την δράση επί της επικουρικότητας των κοινοβουλίων των κρατών μελών. Αν θέλουν να ελέγξουν αυτά τα οποία κάνουμε στο, κοινο, στο νομοθετικό ίτερ, τότε θα πρέπει να το κάνουν μέσω του Συμβουλίου που είναι οι κυβερνήσεις τις οποίες ελέγχουν στη χώρα τους. Η κυρία Γκρέσλε, σας ευχαριστώ για το σημερινό απόγευμα και μιλούσατε για συγκεκριμένες αρμοδιότητες εσωτερική, ε, για παράδειγμα δυνατότητα ελέγχου, το οποίο συγκαταλέγεται στο χαρτοφυλλοκία σας. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία και να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του ελεγκτικού αυτού σκέλους και θα πρέπει να θέσετε λοιπόν τα, τις δικές σας προτεραιότητες. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και δεύτερη ερώτηση, θα δημιουργήσετε και ένα πάνελ ε, ε, ελεγχού και θα καλέσετε τους συναδέλφους σας από την Επιτροπή να κοιτάξετε και να συζητήσουν μαζί σας τα αποτελέσματα του ιστορικού αυτού ελέγχου για να μην μπορείτε να τους εξαναγκάσετε. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξαιρετικά άτομα στους κόλπους της και έχω γνωρίσει ήδη κάποια από αυτά. Έχω εντυπωσιαστεί ιδιαιτέρως ε, και ιδιαιτέρως έχω εντυπωσιαστεί από τα άτομα που εργάζονται σε αυτές τις υπηρεσίες ελέγχου. Είναι πραγματικά πολύ υψηλού κύρους και θα εκτελέσουν με εξαιρετικό τρόπο την εργασία τους και στο μέλλον. Ε, εγώ σας διαβεβαιώνω ότι θα υπάρξει απόλυτη ανεξαρτησία του σκέλους αυτού του ελέγχου, γιατί οι δάλος δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Θα φροντίσω επίσης να ελέγχουν πιο πολύ το output. Αυτό που ε, χορηγείται δηλαδή, κατά πόσον ε, ανταποκρίνεται σε αυτό που περιμένουμε. Αποτελεί το 40% του συνολικού εργασία σήμερα, αλλά θα πρέπει να αποτελέσει μεγαλύτερο ποσοστό για να βελτιωθεί η εργασία μας. Και πιστεύω ότι αυτές οι υπηρεσίε ελέγχου αυτές οι ηλεκτρικές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι ακόμα πιο ανεξάρτητες από τη γενική τους διεύθυνση, προκειμένου να μην υπάρχει η παραμικρή παρέμβαση σε ό,τι αφορά τις κρίσεις τους και τις συστάσεις τους. Και θα ήθελα να πω το εξής. Αν υπάρχουν συστάσεις οι οποίες έχουν εφαρμοστεί ή όχι, μπορείτε ως Κοινοβούλιο να ελέγχετε το τι, ποια ήταν η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζω να το κάνετε αυτό, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ανταπόκριση στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι, λοιπόν, θα φροντίσω οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι αρμόδιοι για θέματα στα οποία έχουν γίνει συστάσεις από τις ελεκτικέ υπηρεσίες να συνεργαστούν μαζί μου προκειμένου στο 100% να εφαρμοστούν αυτές οι συστάσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τίμερμαντς, ο κύριος Νεγκρέσκου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Τίμερμαντς, για να βελτιωθεί η διαδικασία νομοθεσίας γίνεται μία ε, με αξιολόγηση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του πώς ε, γίνεται κάθε φορά η μελέτη αντικτύπου και έχει δεσμευτεί προκειμένου μέχρι τα τέλη του 2014 να δημοσιευτούν νέοι κανόνε. Ένα από τα προβλήματα τα οποία είχαν παρουσιαστεί στα παρελθόν ήταν η διαφάνεια, μάλλον η έλλειψη διαφάνεια. Πότε, θα γίνουν, πότε έγιναν λοιπόν οι μελέτε αντικτύπου και υπό ποιου όρους. Μπορείτε λοιπόν να μα εξηγήσετε ποια είναι η άποψή σα για το πώ θέλετε να βελτιωθεί η διαδικασία αυτή πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις και πώς γίνονται ή θα έπρεπε να γίνονται οι μελέτες αντικτύπου και ε, θέλετε να διαχωριστεί αυτή η διαδικασία από την συλλογή δεδομένων, από την αξιολόγηση ανάλογα με την πολιτική βούληση που ε, υπάρχει. Θεωρώ λοιπόν ως Ρουμάνος ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η διαφάνεια σε ό,τι αφορά το Σέγγεν, σε ό,τι αφορά την διαρτικά ταμεία ή και άλλους πόρους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε, οι μελέτες αντικτύπου δεν είναι εκφύσεως η πρώτη παρότριση, η πρώτη, αν θέλετε, τάση μιας ε, διακυβέρνησης που θέλει να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών του. Δεν τάση, λοιπόν στις μέρες του δικτύπου την πλήρη μου προσοχή και την πολιτική μου προσοχή, θα διασφαλίσω ότι οι υπηρεσίε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα γνωρίζουν ότι θα πρέπει να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να είναι ε, το δυνατόν καλύτερες αυτές οι μελέτες αντικτύπου και μετά θα περάσουν από ε, εξέταση από το σχετικό σώμα μελετών αντικτύπου και θα φροντίσω η σύνθεση των ε, πάνελ αυτών να είναι ανάλογη προκειμένου να υπάρχει σωστή αξιολόγηση, επακριβέστατη. Περίπου το ίμιση των συστάσεων αυτών, των διαπιστώσεων, αποστέλλονται και πάλι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αλλαγή. Και είμαι πεπισμένο ότι έτσι θα πετύχουμε περισσότερα αποτελέσματα. Τούτου λεχθέντος, το ξελέω και το ξαναλέω, αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι τα κοιτάζει αυτά στη φάση που καταρτίζεται η νομοθεσία, αλλά θα πρέπει να το κάνουμε σε όλη τη διαδικασία, στην πρώτη ανάγνωση, στη δεύτερη ανάγνωση, ε, να δούμε τι συμβαίνει στο Κοινοβούλιο, τι συμβαίνει στο Συμβούλιο. Όλα αυτά θα πρέπει να εξετάζονται στα πλαίσια της μελέτης αντικτύπου, γιατί πολύ συχνά αυτό που έχει αρνητικό αντίκτυπο για τους πολίτες, για τις επιχειρήσεις, είναι αυτό που συμβαίνει στην πολιτική διαβούλευση, στο lobbying από τις ε, ομάδες συμφερόντων. Έτσι αλλάζουν οι προτάσει, ακόμα και η ίδια η φύση των προτάσεων. Πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και πρέπει και τα τρία θεσμικά όργανα που συνομοθετούν να αναλαμβάνουν τι ευθύνε του σε ό,τι αφορά τη μελέτη αντικτύπου. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε αυτά λοιπόν μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να βάλουμε και το Συμβούλιο στον αγώνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταία ερώτηση, κυρίε και κύριοι, από την κυρία Γκάλ. Μισό λεπτό, κυρία Γκάλ. Τίμερμανς, μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτηση αυτή μέσα σε δύο λεπτά όπως όλες οι υπόλοιπες και στη συνέχεια έχετε στη διάθεσή σας, αν το επιθυμείτε, πέντε λεπτά για να κάνετε καταληκτικά σχόλια, τα οποία μπορείτε να τα κάνετε κατευθείαν μετά την απάντηση της ερώτησης της κυρίας Γκάλ. Πέντε λεπτά λοιπόν. Κύριε Τίμερμανς, και εγώ η ίδια διαπίστωσα σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αδιαφόρησε. Χαίρομαι ε, που λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα υποχωρήσει στα πλαίσια της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά αυτό θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές εκτιμήσεις και μελέτες. Σαν παράδειγμα, φέρνω τον πίνακα επιδόσεων στον τομέα της δικαιοσύνης. Αναφερθήκατε συχνά στην Ουγγαρία σήμερα και η ανεξαρτησία α, της δικαιοσύνης έχει ανέβει κατά 6 βαθμούς σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Η εμπιστοσύνη στην δικαστική εξουσία είναι περίπου στο επίπεδο που είναι και στη Γαλλία. Αυτό σημαίνει ότι οι αντικειμενικές αναλύσεις δίνουν διαφορετικές εικόνες σε σχέση με τις αναλυθείς αδικαιολόγητες κατηγορίες. Θα μπορέσετε να αναλάβετε την υποχρέωση να παρακολουθήσετε όλα τα κράτη-μέλη με αντικειμενικό τρόπο και θα προστατεύσετε αυτούς οι οποίοι γίνονται ε, αντικείμενο επιθέσεων αδίκως και χωρίς λόγο. Κοιτάξτε, ο χειρότερος εχθρός της, ε, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δικαιωμανάτων είναι ε, η λογική του δεν τρέχει τίποτα. Και εγώ το έχω ζήσει αυτό και ε, στις συζητήσεις που είχα με τον κύριο Λαυρόφ. Όταν έλεγα κάτι για την κατάσταση ε, στην Ρωσία μου απαντούσε άλλα τα άλλων λέγοντας ότι και εσείς τι κάνετε στη χώρα σας γι' αυτό και στην άλλη χώρα τι κάνουν αυτοί γι' αυτό. Ο μοναδικός τρόπος για να διορθώσει κανείς το πρόβλημα είναι πράγματι να μην συγκεντρώνει την προσοχή του μόνο σε μία χώρα και σε μία κατάσταση. Ο μοναδικός τρόπος για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ένωση είναι να είμαστε πλήρως δίκαιοι και αντικειμενικοί για την κατάσταση των κρατών μελών που υφίστανται τον έλεγχο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι τα δεδομένα και τα γεγονότα. Θα το πω και κατά πρόσωπον στον κύριο Ορμπάν. Αν έχω να σχολιάσω μαζί του όσα λέγονται για τη χώρα του και για αυτόν, θέλω πάρα πολύ δουλειά. Αλλά και στην περίπτωση της Ουγγαρίας και στις άλλες περιπτώσεις, εμείς εξετάζουμε προσεκτικά τις λεπτομέρειες. Βλέπουμε ποια είναι τα προβλήματα, ποια είναι τα παράπονα, ποιες είναι οι αναφορές μιλάμε με τους εκπροσώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων, μιλάμε με τους εκπροσώπους του τύπου και τότε διαμορφώνουμε αντίληψη και εικόνα. Και δεν απαντάμε εμείς ε, ε, ότι «Α, εντάξει, εδώ γίνεται αυτό κακό είναι, αλλά αλλού είναι χειρότερο, οπότε δεν ασχολούμαστε με αυτό». Λοιπόν, ε, πρέπει να είναι κανείς δίκαιος και εξαντλητικός. Τώρα, ε, έτσι και αλλιώς πάντα θα μας κατηγορήσουν βέβαια ότι δεν είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί. Αλλά θα πρέπει η κριτική αυτή να φροντίσουμε να μην είναι τεκμηριωμένη και να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι δεν είναι αληθείς οι κατηγορίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απάντησα στην τελευταία υποθέτω ερώτηση και δεν θα σας καθυστερήσω πολύ περισσότερο στα συμπεράσματά μου. Θέλω απλά να μοιραστώ μαζί σας ε, μια αίσθηση κατεπήγοντος θα έλεγα για τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε τα επόμενα πέντε χρόνια. Είμαι πεπισμένος ότι αν αποτύχουμε στα επόμενα δύο χρόνια να συνδεθούμε εκ νέου με τους πολίτες για τους οποίους βρισκόμαστε εδώ, τους Ευρωπαίους πολίτες δηλαδή, τότε το πρόγραμμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης θα απειληθεί εάν δεν συνδεθούμε εκ νέου με αυτούς που λέμε ότι εκπροσωπούμε. Τότε θα γυρίσουν την πλάτη τους ε, στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα και μάλιστα ο άνθρωπος την έφτιαξε καλά την Ευρώπη. Είναι ε, θα έλεγα η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα από τα καλύτερα προγράμματα και σχέδια ειρηνικής συνύπαρξης στον κόσμο. Και όταν λέω την έφτιαξαν ε, οι άνθρωποι εννοώ, δεν εννοώ άνδρες ή γυναίκες. Η γυναίκα μου άλλωστε λέει για να με πειράξει ότι όταν ε, ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, ο Θεός ήταν γυναίκα. Εν πάση περιπτώσει, η επιτυχία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ήταν μεγάλη και δεν θα πρέπει να πάμε πίσω, δεν θα πρέπει να υπαναχωρήσουμε. Και έχω την αίσθηση τα τελευταία χρόνια, βλέποντας και τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα και η Ευρώπη σήμερα, αυτή η τεράστια οικονομική κρίση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε από τη δεκαετία του 30 αυτή η ανυπόφορη αίσθηση απειλής από το εξωτερικό, είτε από τον υπερεθνικισμό της Ρωσίας, είτε από τον ακεραιοφρονισμό στον αραβικό κόσμο. Όλα αυτά δείχνουν δύσκολες στιγμές, για πρώτη φορά μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ε, οι γονείς φοβούνται για το μέλλον των παιδιών τους. Δεν υπάρχουν εθνικές απαντήσεις σε αυτές τις απειλές και σε αυτή την αίσθηση. Απαιτείται μια ευρωπαϊκή απάντηση. Πρέπει όμως για να το κάνουμε αυτό αποδεικνύοντας ότι είναι προς το συμφέρον του Ευρωπαίου πολίτη. Ίσως να θεωρείτε ότι το χαρτοφυλάκιό μου είναι τεχνικής φύσεως. Όμως το να υπάρξουν πιο θετικά και χρήσιμα αποτελέσματα σε επίπεδο νομοθετικό για τον Ευρωπαίο πολίτη είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξανασυνδεθούμε με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των οποίων το μέλλον είναι εν μέρη και στα χέρια μας. Πρέπει λοιπόν να οργανωθούμε σωστά και σε υπηρετικό θα έλεγα επίπεδο, σε κοινοτικό επίπεδο, σεβόμενος τις εθνικές διαστάσεις βέβαια, που συμπεριέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά αν δεν αλλάξουμε τη στάση μας ε, τα επόμενα χρόνια και αν δεν ε, καθορίσουμε σωστά τις προτεραιότητές μας, οι οργανώσεις μας, οι οργανισμοί μας ε, δεν θα έχουν και πάρα πολύ μεγάλο νόημα πια για τον Ευρωπαίο πολίτη. Αυτό δεν θα αφήσουμε να συμβεί. Γιατί αν έχει ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό η Ευρώπη περισσότερο από όλες τις άλλες υπήρους είναι η δυνατότητα προσαρμογής στις νέες προκλήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι θα προσαρμοστούμε, θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και θα πούμε σε λίγα χρόνια στα παιδιά μας ότι σας δίνουμε την Ευρώπη σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι τη βρήκαμε πριν 10 χρόνια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τιμέμαντς ε, και για το ότι κρατήσατε το χρόνο σας. Τώρα, ε, τα μέλη της Επιτροπής της Διάσκεψης των Πρόεδρων που θα ε, κάνουν την αξιολόγηση θα συναντούμε στις 6 ώρα.